Καλημέρα σας. Έχουμε δύο τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη. Η πρώτη φορά την κατάσταση στη Γάζα και τη δράση του Ισραήλ τη Δευτέρα κατά το, της νεοπομπής που κατευθυνόταν στη Γάζα. Ξέρετε ότι πολλοί μεταξύ των οποίων και εγώ, επισκεφθήκαμε τη Γάζα μέσα στα πλαίσια της κοινή ε, επίσκεψης των ε, Επιτροπών ΑΦΕΤ και Budget, έτσι ώστε να δούμε πώς έχει η κατάσταση υπό το φως των διαπιστώσεων μας. Γι' αυτό πρότεινα να ε, συμπληρώσουμε την ημερήσια διάταξη με ένα σημείο που αφορά τις εξελίξεις, πρόσφατες εξελίξεις στην ανθρωπιστική βοήθεια και κρίση στη λωρίδα της ε, Γάζας. Το θέμα αυτό ο, μάλλον ο εκπρόσωπος της Ούνρα στις Βρυξέλλες, ο κύριος ε, Ματίας Μπουσάρ, θα μας ε, πληροφορήσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, έχουμε λάβει δύο ερωτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ώρα των ερωτήσεων και θα πρότεινα να τις δούμε μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης της Συμφωνίας του Κοτονού. Δέχεστε αυτή την τροποποίηση. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ως προς τις τροποποιήσεις της ημερήσια διάταξης όπως έχουν προταθεί. Άρα εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους του Bundestag από, την, από το, τους πράσινους. Τους τρεις εκπροσώπους καθώς και τους ε, βοηθούς τους που θα παρευρεθούν στη συνάντησή μας σήμερα στα πλαίσια ε, ημερίδων μελέτης στο Βέλγιο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσεις. maintenant euh, euh, Αρχίζουμε με τις ε, ανταλλαγές απόψεων με τον Επίτροπο με μεγάλη μας ε, χαρά καλωσορίζουμε τον Επίτροπο υπεύθυνο για θέματα ανάπτυξης, τον Επίτροπο Πιμπάλξ, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τις αναπτυξιακές εργασίες για το 2011. Θα ήθελα όμως ε, πρώτα να συμμετάσχει σε μία απονομή που θα γίνει ε, τώρα Όπως ξέρετε, ήρθα σε επαφή με μη κυβερνητικέ από την Ευρώπη και αφρικανικές οργανώσεις που μου υπέβαλαν μία αίτηση έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τη γεωργία στις χώρες του Νότου. Ορισμένες μη κυβερνητικέ είναι μεταξύ μας και θα τους δώσω το λόγο για τρία λεπτά στην καθεμία έτσι ώστε να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς έχει το ε, διάπημά τους. Δίνω το, το λόγο στην κυρία Πισότ από την SOS και έναν άλλον εκπρόσωπο από την Αγροτική Ένωση του Μαλή. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Πρόεδρε, καλημέρα. Εκπροσωπώ την ε, κυρία Πίσω, τον κύριο Σισοκό. Έχουν πρόβλημα, δεν έχουν ε, μπάτς για να μπουν στο κτίριο, οπότε θα μιλήσω εγώ στη θέση τους. Ευχαριστούμε για την σημερινή σας πρόσκληση. Μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε εξ ονόματος 10 ε, οργανώσεων που εκπροσωπούν την Τσεχία, την Πολωνία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Λουξεμβρού και φυσικά το Βέλγιο. Όλες αυτές οι ευρωπαϊκές οργανώσεις συνεργάζονται με οργανώσεις αγροτών. Θέλουμε να τονίσουμε ότι στην τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιστημιστική ασφάλεια αφορούν στους εταίρους μας για τη συμμετοχή των, της κοινωνίας των πολιτών και των αγροτών ε, για την εμπλοκή τους για τη διαμόρφωση της ε, γεωργικής πολιτικής αυτή η ανακοίνωση λοιπόν μας ε, ικανοποιήσει και θα θέλαμε μαζί με τις οργανώσεις που εκπροσωπούμε να υποβάλουμε κάποια αιτήματα σε σχέση με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Η πρώτη σύσταση που κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε μια πραγματική ουσιαστική εταιρική σχέση με αυτές τις οργανώσεις. Ε, θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματο του κυρίου Σαλή Σοσκό. Σα είπα ότι δεν μπορούσε να μπει στο κτίριο, έχει κάποια προβλήματα. Έχει προετοιμάσει την παρέμβασή του, την έχω γραπτό, οπότε θα σα τη διαβάσω για να καταγράψετε τις προτάσεις του. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε που μας καλέσατε σήμερα. Έρχομαι από το Μαλί και εκπροσωπώ οργανώσεις από την Δυτική Αφρική. Οι προτάσεις που μας υποβάλλουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις σήμερα ε, είναι οι προτάσεις που είχαμε υποβάλει εμείς ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό οι οργανώσεις μας ε, που συμμετέχουν ενεργά στο γεωργικό τομέα θέλουν να συμμετάσχουν στον προσδιορισμό και την υλοποίηση ε, των πολιτικών στήριξης της γεωργίας στις χώρες μας. Επίσης, εδώ και πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών, με τις ε, χώρες του Νότου για να υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια πρόσφατη ανακοίνωσή της επανέλαβε τη δέσμευσή της και επίσης έκανε αντίστοιχη δήλωση το Συμβούλιο. Επιτόπου δυστυχώς δεν έχει σημειωθεί καμία αλλαγή. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, στο Μαλί, παραδείγματο χάρη, ε, είχαμε 33 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν σε ένα πρόγραμμα επιστημιστική ευαισθητοποίησης και σε ένα πρόγραμμα της Παγκόσμια Τράπεζας, χωρίς όμως πρώτερη διαβούλευση με τις οργανώσεις μας. Ο αντίκτυπος ε, για, για το γεωργικό δυναμικό της χώρας μας ήταν αμεληταίο. Οπότε θα θέλαμε να το λάβετε υπόψη σα και μαζί με τι ευρωπαϊκέ οργανώσει προτείνουμε προτείνουμε το εξής. Τις ερχόμενες εβδομάδες να διοργανώσουμε μία συνάντηση ανάμεσα στη δική σας διοίκηση και τους εκπροσώπους των οργανώσεων της Δυτική Αφρικής, ούτω ώστε να συμφωνήσουμε σε επισκεκριμένων όρων για την υλοποίηση της πολιτικής στήριξη της γεωργικής παραγωγής στι χώρε μας. Στην Δυτική Αφρική ξέρετε ότι έχουμε και σε περιφερειακό επίπεδο πολιτικές και σε διεθνικό Υπάρχει κοινή οργάνωση και υπάρχει ενεργό συμμετοχή για τον προσδιορισμό των πολιτικών που εφαρμόζεται στις διάφορες χώρες. Ας εργαστούμε μαζί και ας αρχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ας μην ξεχνάμε τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, διότι θέλουμε να δώσει τα αποτελέσματα αυτή η συνεργασία μας, το ταχύτερο δυνατόν. Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών στήριξη τη γεωργίας θα επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία των αγροτών και των οργανώσεών του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτό το σημαντικό μήνυμα. Τώρα θα υποβάλω αυτό το αίτημα στον Επίτροπο Πίμπαλξ. Il faut prendre en considération leurs <clears throat> observations et revendications. Donc, Για να ε, γυρίσουμε τώρα ε, στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή στο διαρθρωμένο διάλογο για τις προτεραιότητες της Επιτροπής το 2011. Ο κύριος Ελένε στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών κάλεσε τον Επίτροπο για το διαρθρωμένο ετήσιο διάλογο, ούτω ώστε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες νομοθετικές προτεραιότητες απαραίτητες, οποίες θα κοινοποιήσουμε στη συνέχεια στον κύριο Λένε θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 και όχι για το 2010 που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2010. Ο στόχος συζήτηση με τον Επίτροπο είναι μεταξύ άλλων να του δώσουμε την ευκαιρία να μοιραστεί μαζί μας κάποιες από τις προθέσεις του για το 2011 και έτσι να συμβάλλουμε και εμείς στο χρονοδιάγραμμα εργασιών για το 2011, διότι θα το αναφέρουμε τις δικές μας προτεραιότητες και τις ενδεχόμενε ατέλειες που θα εντοπίσουμε στο ε, ανακοινωθέν πρόγραμμα της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, εξέτοιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, είναι, έχουν πέρασει 50 χρόνια από την δημιουργία των πρώτων σχέσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και των αναπτυσσόμενων χωρών στην αρχική συνθήκη της Ρώμης, δηλαδή πέντε δεκαετίες ανάπτυξης. 50 χρόνια πριν η... διακηρύχθηκε η μέρα της ανεξαρτησίας για την Αφρικανική Ήπειρο έτσι ώστε η χώρα να μετατραπεί σε αυτό που, ξέρουμε, που γνωρίζουμε σήμερα. Και έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από τη δημοσίευση της, ε, της τελευταίας έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας που πρότεινε πρώτη έναν στόχο ε, βοήθειας για τον αναπτυσσόμενο κόσμο του 0,7% του ε, ακαθάριστου ε, χώρου προϊόντος. Μέχρι το 1975 είχαμε θέσει ένα στόχο ο οποίος ε, θα τρέχει μέχρι το 2015. Στην πολιτική αυτή ο χρόνος περνά γρήγορα και δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Είμαστε ήδη στο 2010 και είναι πραγματικά ο χρόνος κλειδί για την ανάπτυξη. Όπω είπα στην ακρόασή μου ενώπιον αυτή τη επιτροπή, είμαι επεπισμένος και θέλω να κάνω ε, την αλλαγή στην ε, άρση της φτώχεια φτώχειας ε, κατά τη διάρκεια τη θετίας μου στι πιο φτωχέ περιοχέ. Ο βασικό μου στόχο λοιπόν είναι να καθορίσω τις ε, προοπτικέ για μια νέα δεκαετία για την ανάπτυξη. Θέλω να χαλκεύσω μια σημαντική σχέση με την Επιτροπή αυτή, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανάπτυξη να είναι μια πολιτική περηφάνεια για όλου μα. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τομεί, αλλά η ανάπτυξη δείχνει τι κοινέ αξίε που μοιράζεται η Ευρώπη και την κοινή διάθεση που υπάρχει για να τι εφαρμόσουμε αποτελεσματικά. Καθόρισα το όραμά μου σε μια επιστολή που σα είχα στείλει την προηγούμενη εβδομάδα και υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι γιατί πιστεύω ότι μπορούμε όντως να κάνουμε τη διαφορά. Εξακολουθώ να, το 2010 να το θεωρώ ένα έτος ευκαιρίας. Εξακολουθώ να χαίρομαι όταν αναφέρω τους πιο, τα βασικά ορόσημα τα οποία θέλω να επιτύχω φέτος. Η πρώτη ευκαιρία είναι η νέα, μια νέα αναπτυξιακή πολιτική και το σχετικό πλαίσιο από, τα, από, την, από την συνθήκη της Λισαβόνας. Με την δράση μας και με την μακροπρόθεσμη, ε, η, η δράση μας σε ό,τι αφορά την, την άρση της ε, της φτώχειας είναι μια από, ένας από τους βασικούς μας στόχους. Και βεβαίω αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στα πλαίσια των εξωτερικών δράσεων παγκοσμίω. Για να... Ήδη του ή το θέμα της ε, απαλήψη της φτώχεια έχει μπει και στους στόχου τη χιλιετίας και εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε εάν έχουμε το πολιτικό θάρρο η πρόοδος που έχει γίνει είναι καλή έτσι ώστε να μειώσουμε όντως τη φτώχεια. Αλλά το θετικό, ένα θετικό μήνυμα δεν σημαίνει τίποτα αν είσαι ένας από τους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των στόχων της χιλιετίας, τα κράτη-μέλη έχουν υποσχεθεί να αυξήσουν τη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες η δική μας πρόκληση είναι να πείσουμε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν ε, την ε, αναπτυξιακή βοήθεια ακόμη περισσότερο. Οι Ευρωπαίοι έχουν δεσμευθεί και δείχνουν ε, υποστήριξη για την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό φαίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρά τις οικονομικές δυνατότητε, αυτό ούτε τα τελευταία χρόνια. Τις οικονομικές, τα οικονομικά προβλήματα ούτε τα τελευταία χρόνια άλλαξε αυτό. Ελπίζω λοιπόν να μπορώ να, στηριχθώ και στην δική σας στήριξη και στις, ε, τη στήριξη των ε, ε πρωτευουσών της Ευρώπης. Το να τηρήσουμε τις ε, ε υποσχέσεις μας δεν, είναι απλώς, δεν πρέπει να είναι απλώς εφικτό, αλλά πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος. Έχουμε τις κλιματικές αλλαγές, ένα μακροχρόνιο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει κυρίως αυτούς που δεν φταίνε. Επίσης ε, είναι προς το συμφέρον μας να βοηθήσουμε, όχι μόνο ηθικά, αλλά να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια για τους πολίτες μας και να προωθήσουμε την, κοινωνική, την οικονομική ανάπτυξη. Εγώ θα ήθελα να, ε, να βασίσουμε αυτές τις υποσχέσεις σε επιτυχίες. Θέλω να κάνουμε τη διαφορά, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ των Ευρωπαίων φορολογουμένων θα δαπανάτε, που δαπανάτε θα έχει και αντίκρισμα. Αυτό ε, πρέπει να, αυτό πρέπει να δούμε πώς, γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα μόχλευσης ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Σημαίνει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις, ε, στη βοήθεια που δίνεται στις ε, περιοχές που όντως υπάρχει ε, δυνατότητα να δράσουμε εμείς σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να ξεπεράσουμε απλώς τα, τα, τα, νούμερα και να δούμε την πραγματική επιρροή που μπορεί να έχει ανάπτυξη, στην ανάπτυξη στην επιστηστική ασφάλεια, στις ε, θέσεις εργασίας, ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών που, των αναπτυσσομένων. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, δείχνοντας επίσης και πώς η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να καταστήσει πιο αποτελεσματική την αναπτυξιακή βοήθεια, εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει διαβούλευση μεταξύ της Κομισιόν και των 27 κρατομελών, καθώ επίση και συντονισμό. Μπορούμε έτσι να έχουμε μεγαλύτερη ε, αξία, να έχουν τα χρήματα που δίνουμε μεγαλύτερη αξία. Θέλω όντω να προχωρήσουμε πραγματικά ώστε να έχουμε ένα έγγραφο ε, ε, κοινοτικό για κάθε χώρα που θα λάβει την αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης ε, θέλω να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μας μέσω συνακτικής πολιτικής. Η, ε, επιρροή που μπορούν να έχουν οι πολιτικές αυτές στην, ε, στις, στις χώρες αυτές ε, είναι σημαντικές. και η αύξηση του ΑΕΠ είναι επίσης πολύ σημαντική. ο συντονισμός, η διαβούλευση και η, συμπληρωματικότητα, όλα αυτά απορρέουν από τη νέα συνθήκη η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει το εργαλείο ώστε να κάνουμε την ε, ελπίδα προσδοκία. Την ελπίδα μας να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια στην προοπτική μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής η οποία θα επιτύχει τους στόχους της χιλιετίας έτσι ώστε η ε, βοήθεια να γίνει ε, μια προοπτική συντονισμένης απάντησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι επίσης οι, οι πολιτικές μας δεν θα βλάψουν την, ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ο δεύτερος λόγος γιατί είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε όντω να κάνουμε την διαφορά είναι η εταιρική μας σχέση με την Αφρική. Οι σχέσεις ε, Ήπειρο με Ήπειρο που έχουμε με την ε, Αφρική είναι μοναδική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει ένα πλαίσιο το οποίο ξεπερνά την, ε, τη σχέση δωρητή και λήπτη, αλλά δημιουργεί ίσους ε, εταίρους ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για να επιτευχθούν οι στόχοι της ε, χιλιετίας, να προωθήσουμε την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, οι σχέσεις μας με την Αφρική ξεπερνούν την ανάπτυξη ώστε να μπορούμε να, να συζητούμε την ασφάλεια, την ειρήνη, τα δικαιώματα, την διαφάνεια και την... τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφάνεια και την πρόσβαση. Και εγώ θέλω ότι αυτή η βοήθεια να αποτελέσει τον καταλήτη προς την καλή διακυβέρνηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα ότι χωρίς καλή διακυβέρνηση η ε, προσπάθειά μας δεν θα έχει αποτελέσματα και σε, περιπτέ... σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και αντιπαραγωγική, ειδικά σε ό,τι αφορά τις χώρες που είναι πλούσιες σε πόρους. Is Επίσης, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς ε, τομείς και μία από τις βασικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και ο αναπτυσσόμενο κόσμο είναι αυτό που επηρεάζεται περισσότερο. Επίσης, ως στον αναπτυσσόμενο κόσμο και ειδικά στην υποσαχαρία Αφρική αναμένεται από, το από, τον, από τον ΟΗΕ να αποτελέσουν τα μέρη αυτά ε, μία από τους, ε, από τους βασικούς παίκτες στην, στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Είναι λοιπόν μεγάλες οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε, σε ό,τι αφορά και τις εκπομπές του εξουδίου του άνθρακα για αυτές τις χώρες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλέ θετικέ ευκαιρίε. Ε, στην ε, διάσκεψη τη Κοπεχάγη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να δώσει σημαντική χρηματοδότηση για το, για την, ε, στον αναπτυσσόμενο κόσμο για το Ταμείο τη Παγκοσμιοποίηση. Επίση, η σωστή χρήση των κονδυλίων θα εξασφαλίσει ότι ο αναπτυσσόμενο κόσμο θα έχει τις δυνατότητες που χρειάζεται για ανάπτυξη. Ιδιαίτερα είναι σημαντικό ότι πολλοί, πολλές, πολλές χώρες στον αναπτυσσόμενο χρόνο αποτελούν ε, ε, το καταλληλότερο σημείο για να αναπτυχθούν νέες μορφές ενέργειας. Ηλιακή ενέργεια, ε, αιωλική, υδροηλεκτρική. Σε πολλά μέρη της Αφρικής μπορούν να γίνουν αυτά. Σε, μπορούν να γίνουν λοιπόν επενδύσεις ώστε να παραχθεί με βιώσιμο τρόπο να παραχθούν νέα βιοκαύσιμα. Σε υγεία πούμε που δεν χρησιμοποιείται για ε, τη γεωργία. Ε, συνδυάζοντας λοιπόν και, τα, και την δυνατότητα μόχλευσης αλλά και, την, και τα αναπτυξιακά κονδύλια και χρησιμοποιώντας και τα κονδύλια που έχουμε δώσει ως συνέπεια της ε, Συμφωνίας της Κοπενχάγης μπορούμε όντως να κάνουμε την διαφορά δεδομένου ότι θα έχουμε και την, θα, θα μπορέσουμε να μονώσουμε ουσιαστικά τις χώρες της, του αναπτυσσόμενου κόσμου από την καταστροφή που φέρνουν οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου. Οι χώρες της Αφρικής πρέπει να δράξουν αυτή την ευκαιρία ώστε μέσα από αυτή τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής να δώσουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται σε κάθε πολίτη μέσω των νέων επενδύσεων που θα γίνουν. Η κλιματική αλλαγή και η ανάπτυξη επίσης είναι σημαντική τομή. και μαζί με, τον συνάδελφο Χέντεγκαρτ, με τη συνάδελφο Χέντεγκαρτ ε, έχουμε συνεργαστεί ως προς ε, τον τομέα αυτό οπότε έχουμε πολλούς ε, λόγου για να είμαστε αισιόδοξοι. Την διάσκεψη τη Κοπεχάγη, την βιώσιμη ανάπτυξη και την, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Επίση, τι προτίθεμαι να κάνω, θα σας πω, στους επόμενου μήνε για την κλιματική αλλαγή και για να βοηθήσουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Καταρχήν, θέλω να παρακολουθήσω το σχέδιο δράσης των 12 σημείων που είναι μέσα στους στόχους της χιλιετίας και που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν τον Απρίλιο. Αυτό φαίνεται να είναι το καρμπόν για την ε, για, τον, ε, για τη διάσκεψη κορυφής που θα γίνει τον ε, Σεπτέμβρη και θέλω να εξασφαλίσω τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική υποστήριξη ώστε η Ευρώπη να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο. Θα ευχαριστήσω τον Μέκλ Κάσμαν για την δουλειά που έκανε, για την έκθεση, την οποία ολοκλήρωσε η Επιτροπή σας. Επίσης, δοκιμάσαμε τις ιδέες αυτές και με τους εταίρους μας στην Λατινική Αμερική, την Ασία και την Καραϊβική την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια, μια συνάντηση ε, του Κολεγίου των Επιτρόπων. Εγώ πήγα σε μια διάσκεψη του ΑΣΕΜ ε, πριν από καμιά εβδομάδα, οπότε προσπαθώ να πιέσω και τους υπουργούς στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι το Συμβούλιο Κορυφής της, του Ιουνίου θα πετύχουμε να ενισχύσει τις ιδέες μας, να υποστηρίξει τις ιδέες μας, γιατί αυτή είναι η ερχοκοκαλιά της ε, συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της G8 και της G20 στον Καναδά. Επίσης, νέα φάση στην ε, εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Το Νοέμβρη, στην Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική, θα τεθεί το νέο πρόγραμμα δράση για τι δύο ε, υπήρου τα επόμενα χρόνια. Θέλω αυτό να ξεπεράσει την, ε, το να βασιστούμε μόνο στις παλαιότερες επιτυχίες. Η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής αποτελεί το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,8 ε, ε, δισεκατομμύρια άτομα που, κάθονται, που ουσιαστικά εκπροσωπούνται γύρω από ένα τραπέζι. Θα έχουμε λοιπόν και κατευθυντήρες γραμμές για την, ε, για την ε, κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που θα εκδοθούν ε, αργότερα μέσα στο έτος. Επίσης θα επικεντρωθώ στο πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα ωφέλη από τις νέες εξωτερικές σχέσεις και τις προοπτικές που προκύπτουν και που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και τη νέα ε, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Επίσης ε, πρέπει να πω ότι ούτε η Βαρόνι Άστον ούτε εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια απειλή για την αναπτυξιακή πολιτική. Είναι μια ευκαιρία και ο βασικός μας ε, γενικός στόχος θα είναι αυτός ακριβώς. Αυτή είναι η, αυτός είναι ο βασικός μας στόχος για τις εξωτερικές μας σχέσεις η απάλληψη της φτώχειας είναι το καταλληλότερο όπλο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία, την έλλειψη ασφάλειας, την τρομοκρατία, να, ενισχύσουμε την καλή διακυβέρνηση, τα σοβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δώσουμε την, τα απαραίτητα κονδύλια για την εμπορική ανάπτυξη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι όλα αυτά τα, τα στοιχεία των εξωτερικών μας σχέσεων και της στρατηγικής τους θα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και ότι η, Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα εργαστεί ως ε, μία δύναμη. Εγώ ξεκίνησα με δύο ανακοινώσεις μαζί με τη Βαρονιά Άστον ως προς αυτό, ώστε να έχουμε μία συνεκτική εξωτερική πολιτική, πολιτική εξωτερικών δράσεων και μια αναπτυξιακή ε, πολιτική για το κέρας της Αφρικής και για το Αφγανιστάν. Δεν θα πρέπει να σας εκπληξεί ότι όταν εφαρμόζουμε την ε, ε, το πρόγραμμα αυτό, υποστηρίζοντας και τους ε, στόχους της χιλιετίας, ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα της, ε, του ευαίσθητου χαρακτήρα που υπάρχει στις χώρες αυτές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια που πάνε στις χώρες αυτές θα έχουν όντως αποτέλεσμα και αντίκρισμα. Το δεύτερο μισό λοιπόν του έτους θα εκδώσω μια πράσινη βίβλο για την ε, ε, δημοσιονομική στήριξη, ενίσχυση. Αυτό έχει γίνει, έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Περίπου το μισό των ταμείων Ε, δίδεται από του ε, εθνικού προπολογισμού. Ελπίζω να έχουμε μια ε, καλή ειλικρινή συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ώστε να προσαρμοστεί το εργαλείο αυτό στις νέες εξελίξεις. Φτάνω στα τελευταία μου σχόλια. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή και αυτό φέρνει μαζί του την ανάγκη να αναθεωρήσουμε την συμφωνία που υπήρξε για την, ανάπτυξη, για την ανάπτυξη στα πλαίσια του 2011. Χρειαζόμαστε μια αναπτυξιακή πολιτική που θα είναι προσαρμοσμένη στις νέες πραγματικότητες. Οι χώρες εταίροι σε όλο τον κόσμο έχουν χτυπηθεί πολύ από την ε, οικονομική κρίση. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, πολύ είναι διπλά δύσκολο να ε, κάνουμε πραγματικότητα αυτά που είχαμε υποσχεθεί. Πρέπει λοιπόν να, έχουμε, να προσαρμοστούμε στη νέα γεωπολιτική κατάσταση. Χρειάζεται νέα ε, ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου και την, ε, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάθεσης του Κοινοβουλίου και των Κρετών μελών και θέλουμε η αναπτυξιακή πολιτική να είναι προσαρμοσμένη στη νέα δικαιατία. Να μειώσουμε το, μέχρι το 2015 50% τη φτώχεια παραμένει ένας στόχος ρεαλιστικός. Παρ' όλα αυτά αυτό είναι το εύκολο. Η ε, επάλυψη της φτώχεια που είναι ο, ο τελικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωση θα είναι μεγαλύτερη ε, πρόκληση. Γι' αυτό τώρα προσπαθώ να εκπονήσω την στρατηγική που θα πρέπει να μας απασχολήσει για την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. I will now give the floor to the member. Για αυτή την ανακοίνωση, ο κύριος είναι ο πρώτος ομιλητής, δίνω το λόγο στους ομιλητές. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μεταξύ μας για αυτή την εξαιρετική παρουσία. Είπατε ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι για μας ε, μεγάλη προτεραιότητα, ίσως για όλους εμάς σε αυτή την αίθουσα, αλλά όχι για όλα τα κράτη-μέλη, γιατί η Ιταλία δίνει ένα 0,1% του ΑΕΠ για τις αναπτυξιακές πολιτικές βρισκόμαστε στο κατώτερο σημείο, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν ε, ένα ιστορικό ως προς την αναπτυξιακή πολιτική και ε, βοήθεια. Οι φιλελεύθεροι στην Ολλανδία μιλάνε για μείωση 50% της αναπτυξιακής βοήθειας, ε, ενώ είχαν μια μεγάλη προϊστορία σε αυτό το τομέα. Εμείς από τη δική μας Επιτροπή και εσείς από την Κομισιόν θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη γιατί είναι δύσκολο να κερδίσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο και δεν νομίζω, δεν είναι εύκολο να φτάσουμε σε δεσμευτικές συμφωνίες για να τηρήσουμε το 0,7% του ΑΕΠ. Αυτό δηλαδή το κριτήριο. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες έτσι ώστε η Επιτροπή να εξεύρει τρόπο για δεσμευτικές συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε όλοι να τηρήσουμε το 0,7% του ΑΕΠ. Μας ε, το υποσχέθηκαν ε, μερικά χρόνια πριν, αλλά φαίνεται ότι δεν τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Πέρα από αυτό το θέμα της χρηματοδότησης, πιστεύω ότι ε, έχουμε να κάνουμε με βαθμία ανάπτυξη των ελευθεριών. Και εγώ ήμουν στην Αιθιοπία μερικές βαμάδες όπως και εσείς και οι εκλογές στην Αιθιοπία οποία ε, δεν ε, ανταποκρίθηκαν στις ε, διεθνείς προδιαγραφές δυνάμει του και του αιθιοπικού νόμου. Είναι μια μεγάλη χώρα της Αφρικής, αλλά έχουμε να κάνουμε με μια realpolitik που περιμένουμε πολύ περισσότερα από την Αιθιοπία παρά από την Γουινέα Μπισάου, διότι είναι μία από τις πιο σταθερές χώρες στην περιοχή. Η πολιτική ανάπτυξη απαιτεί κάθε, κάτι περισσότερο από τη Realpolitik. Όχι μόνο μείωση της φτώχειας, αλλά και αμοιβαία αύξηση των ελευθεριών σε μια χώρα όπως η Αιθιοπία έτσι ώστε να προωθήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, την ελευθερία να επιλέξει κανείς τη δική του κυβέρνηση χωρίς ε, δυσκολίες. Καλή διακυβέρνηση, όπως είπατε κι εσείς. Υπ' αυτή την έννοια, θα ήθελα να μας ε, διευκρινίσετε λίγο περισσότερο τις ε, ευθύνες σας στο EAS γιατί η πρόταση όπως είναι διατυπωμένη σήμερα δεν είναι τόσο αποσαφηνισμένη όσο θα θέλαμε εμείς. Έτσι ώστε να μιλάμε για πραγματική ε, ανάπτυξη, δηλαδή όχι μόνο έλλειψη φτώχειας, αλλά και πλήρη ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. ε, πολύ φοβάμαι ότι οι πολιτικές προτεραιότητες θα παραμείνουν στη σφαίρα της realpolitik και όχι στην πραγματοποίηση των ε, αυτών πραγματικών στόχων. Ως προς τη νέα αναπτυξιακή εποχή, εάν μιλάτε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, θα πρέπει να μην μιλάμε για χώρες ΑΚΕ είναι ε, μία μεταπικιακή ε, αντίληψη. Έχουμε διανύσει 50 χρόνια και νομίζω ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτή την επώδυνη μεταπικιακή ιστορία που ίδρυσε τις χώρες και Θα πρέπει να βασιζόμαστε σε μια συλλογιστική του μέλλοντος με χώρες οι οποίες είναι φτωχότερες από τις δικές μας, έχουν χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα, αλλά έτσι να το δούμε το θέμα. Και οι χώρες ΑΚΕ είναι η συνέχεια μιας απολυθωμένης έννοιας. Thank you, Michael. Thank you. παρακαλώ να περιοριστείτε στο χρόνο ομιλίας. Σε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, γιατί είμαι ο πρώτος στον οποίο ισχύει ο περιορισμός του χρόνου ομιλίας, μεγάλη τιμή μου. Θα ήθελα να θίξω ορισμένα θέματα από την παρουσίαση του Επιτρόπου Πιμπάλξ. Ξέρω ότι έχει πολύ καλή, υπάρχει πολύ καλή θέληση. Αλλά θα ήθελα να είμαι προκλητικός. Είπατε ότι εμείς θα κάνουμε τη διαφορά. Αναρωτιέμαι κατά πόσο δεν θα μπορούσε να γίνει μεταξύ αυτού που προανακοινώθηκε και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε για 0,7%. Αυτό ανακοινώθηκε. Αυτό τόνισε και ο προλαλής σας και θα πρέπει να πω ότι η υπόσχεση του 0,7% δεν θα μπορέσει να τηρηθεί γιατί έχει υποτιμηθεί το ευρώ έναντι του δολαρίου. Η Επιτροπή έχει δει ποιε είναι οι επιπτώσεις. Ε, ένας άλλος παράγον είναι το, το χρέος, το οποίο ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με τη μελλοντική του εξέλιξη. Αυτό δεν είναι παρά η βιτρίνα της ουσίας. Το ίδιο ισχύει για την Ισπανία υπάρχει, έχουμε να κάνουμε με μια παρόμοια βάση σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς το ευρωπαϊκό κονσένσου στην Ευρωπαϊκή Συνένωση για την Αναπτυξιακή Πολιτική υπάρχει αυτή η συνένεση από το 2005. Όλοι έχουμε προσχωρήσει σε αυτή τη συνένεση με βάση μια διαπραγμάτευση που έγινε από τον προκάτοχό σας. Είναι μια πολύ καλή βάση με πολύ καλές προβολές για το μέλλον. Τι κρίνεται ότι είναι αναγκαίο έτσι ώστε να γίνει μια αναθεώρηση. Υπάρχουν βασικά στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε συζητήσεις και σε αυτή την περίπτωση θα θέλαμε να ξέρουμε τι σκέφτεσαι, τι σκέφτεστε επ' αυτού. Ως προς τις δημοσιονομικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις και τις ε, οικονομικές ε, δυσκολίες, θα ήθελα να αποτιμήσουμε όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης για να φτάσουμε στους στόχους. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος υπόκειται σε προθεσμίες και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε καταρχήν το AIDS, την ελονοσία, τη φυματίωση. Υπάρχουν ειδικά ταμεία για αυτές τις ανάγκες και νομίζω ότι δεν είμαστε επαρκείς όταν πρόκειται για ε, ανάγκες πολλοένα και πολλαπλασιάζονται και όπου οι Αμερικανοί ζητούν ε, να καταβάλουμε εμείς το 1 τρίτον και γι' αυτό ακριβώς ε, πιστεύω ότι εμείς έχουμε μία ηγετική θέση στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Μιλήσατε για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, τις σχέσεις με την κυρία Άστον Κατά την άποψή μου, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να βρει τις κατάλληλες συνέργειες με βάση τη, τα, τα διαφορετικά συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο οι άλλες συνιστώσεις θα παρέμβουν άμεσα για να ε, βοηθήσουμε σε αυτή την αναπτυξική πορεία. Υπάρχει κάτι που ε, ε, είναι απαγορευτικό, ας πούμε, ως προς αυτή την προθεσμία των πέντε μηνών. Είσαστε ικανοποιημένος ή υπάρχουν προσκόμματα. Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Ο κύριος Κάσμαν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Αρχικά θα ήθελα να πω πως πρέπει να συνεργαστούμε. Αλλιώς η ανάπτυξη και όλες οι αρχές που υποστηρίζουμε μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα στεφθούν με επιτυχία. Είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε. Ξέρω ότι ανησυχούν όλοι για την έκβαση των διαπραγματεύσεων Κοτονού. Θα τα πούμε αργότερα. Προς το παρόν, να σας πω, Επίτροπε, ότι δεν αμφισβητώ τη δέσμευσή σα για την υπεράσπιση των θεμελιωδών ε, ελευθεριών, των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και την ε, προστασία κατά της ελονοσία, ε, του AIDS και την προστασία όλων των φιλομεταβατικών, ομοφιλοφίλων, αμφιφιλοφίλων κτλ. Αλλά ξέρετε, δεν μπορείτε να ιεραρχήσετε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμεί τα δικαιώματα σε κάποιε χώρε. Είναι οικουμενικά και ούτω ή άλλω είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των χωρών. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προάγουμε, να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα στο Μαλάουι, στην Κένια, σε άλλες χώρες. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, υπάρχει φτώχεια και προσπαθούν όλοι να βρουν έναν αποδιοπομπέα τράγο και αυτό το βλέπουμε στις καταδιώξεις των κοινοτήτων των ομοφιλοφίλων. Πρέπει να βρούμε και άλλα μέσα και άλλα εργαλεία για να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες όλων ε, στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας. Η βιωσιμότητα ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντική όπως και η βιωσιμότητα στην οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τα δικαιώματα, να τα υποστηρίξουμε και να τα προαγάγουμε. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Η έκθεση των στόχων της χιλιετίας απηχεί, ξέρετε, τη θέση της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής. Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες για την υποστήριξή τους. Καλωσορίσουμε το σχέδιο δράσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο, αλλά ξέρετε, οφείλω να πω επίσης ότι δεν με εμπνέει η θέση που τώρα εκπονείται στο Συμβούλιο. Ε, δεν υπάρχει ηγεσία, δεν υπάρχουν νέες δεσμεύσεις, ε, δεν έχει καμία σπίθα, καμία ζωή. Τέλος, και θα κλείσω και την παρέμβασή μου, Πρόεδρε, για την κατάργηση της πολιτικής ΑΚΕ δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Νόμιζα ότι υπήρχαν προβλήματα, αλλά ότι, εν πάση περιπτώσει, ήταν ο τρόπος για να ξεπεράσουμε το κρατικό παρελθόν μας. Αλλά ίσως ο, να τα με τον Τάισον πριν επιβάλλουμε τις απόψεις μας σε άλλους. Ξέρετε, Πρόεδρε, δεν, ε, είναι παράλογο για μένα όταν ε, τη της οικονομικής ε, παγκόσμιας κρίσης ε, να αποσυρθούμε, να επαναχωρήσουμε από τις δεσμεύσεις μας για οποιαδήποτε χώρα. Τους έχουμε ζητήσει να δεσμευθούν για τόσα δις, για ένα ποσοστό του ΑΕΠ τους, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους. εντάξει, μπορεί να είναι χαμηλό γιατί έχουν δυσκολίες, αλλά θα κατανεμηθούν λιγότερα κονδύλια. Αλλά τι, να αποσυρθούμε τώρα σε τόσο κεντρική στιγμή. Συγγνώμη, αν το κάνουμε αυτό τώρα, θα, σαν τον Κράτσο Μάρξ θα καταλήξουμε. Δηλαδή θα λέμε έχουμε αυτές τις αρχές, αλλά τελικά μπορούμε και να τις αλλάξουμε αφού άλλαξαν τα δεδομένα, αφού άλλαξε η κατάσταση. Μα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω κι εγώ για λίγα λεπτά. Euh, Μας μιλήσατε για την ε, συνοχή ανάμεσα στις διάφορες εξωτερικές πολιτικές. Η Επιτροπή Ανάπτυξης από κοινού με την Επιτροπή Αλίας στις 22 Ιουνίου διοργανώνουν από κοινού ένα σεμινάριο. Και έχουμε προσκαλέσει έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που έχει αξιολογήσει τις πολιτικές και τις διάφορες ε, συμφωνίες ε, που έχουμε προσυπογράψει. Έκανα λοιπόν μια ανεξάρτητη αξιολόγηση και τον έχουμε προσκαλέσει ε, σε αυτή την κοινή ακρόαση που διοργανώνουμε. Στη Γάζα δυστυχώς έμαθα ότι η γάμα δέλτα μάρε αρνείται να έρθει ο εμπειρογνώμονας αυτός στη συνεδρίασή μας. Δηλαδή ισχυρίζονται ότι είναι ανάρμοστο να προσκαλούμε εμείς ανεξάρτητο εμπειρογνώμονο που έχει αξιολογήσει ε, αυτές τις συμφωνίες. Κύριε Πίμπαλξ, Ε, μπορείτε να παρέμβετε γιατί είναι απαράδεκτο η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ να μας ε, εμποδίζει να ακούσουμε την ε, αξιολόγηση αυτού των εξάρτητων εμπειρογνώμων για την θαλάσσια πολιτική. Συγγνώμη, αυτό είναι η αγαστή συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Όχι. Νομίζω ότι έτσι προσπαθούν να ελέγξουν τις πληροφορίες. Αν η ΓΑΜΑ ΜΑΡΕ θέλει λοιπόν να ελέγχει τις πληροφορίες, αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία συνοχή ανάμεσα στην αλληλευτική πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Δεν θα το δεχτώ να μας εμποδίσουν να προσκαλέσουμε τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Στην επιστολή που μου στείλατε, λέτε και φυσικά συμφωνώ απολύτω ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να πιέσουν τους πολίτες τους ε, να, ε, ώστε να αρχίσουν να ανεβαίνουν την κλίμακα της ανάπτυξης. Αυτό δεν κάνουμε, αυτό κάνουμε, συμφωνούμε απολύτως. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επενδύσει 48 εκατομμύρια ευρώ στο ε, ορυχείο Κομπάνι που ανήκει στην Glencore που είχε το αρχηγείο της στην Ελβετία. Δεν έχουν πληρώσει ποτέ φόρους λοιπόν. Και γιατί έγινε αυτή η επένδυση για να χρησιμοποιήσουν οξύ, για να βγάλουν το χαλκό από το ρηχείο. Αυτό ε, είχε ως αποτέλεσμα πολλά ατυχήματα. Το φορολογικό καθεστώς δίνει μόνο 1% στη Ζάμπια από το εισόδημα, παρότι δηλητηριάζουν τα πάντα, έχουν χείριστες συνθήκες εργασίας, προκαλούν ατυχήματα με τη μέθοδό τους. Τι προτείνετε να κάνουμε για αυτές τις επενδύσεις ε, που γίνονται για να ε, λαμβάνει περισσότερα χρήματα τουλάχιστον η Ζάμπια. Στην επιστολή σας επίσης είπατε ότι θέλετε να υπάρχει μια ενοποιημένη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια, για το κράτος δικαίου, για την καταπολέμηση της πειρατείας, ε, για ολόκληρη την Αφρική. Αυτό συνάδει με τη δική μας άποψη εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης Αυτό είναι πρόδρομος της μελλοντική ε, πολιτικής σας. Ε, θέλω να ρωτήσω, δηλαδή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης αυτό προτίθεται να κάνει, να εκχωρήσει σε εσά όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Και πριν αρχίσουμε δεύτερο γύρο ερωτήσεων, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και όλες τις υπόλοιπες ε, των προλαλισσάντων. Παρακαλώ. Well, thank you, Mrs. Προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Αρχίσουμε με την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο δεσμευτική συμφωνία από το 0,7%. Θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα και η ανάπτυξη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε περικοπή των ε, χρημάτων των κονδυλίων τη στιγμή που υπάρχει προστιθέμενη αξία. Ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο η νέα κυβέρνηση, όχι η παλαιά, αλλά η νέα μπορεί να αφήσει ανέπαφη την παλαιά πολιτική με καλές ε, προθέσεις γιατί οι σωστές πεπιθήσεις οδηγούν στην προστιθέμενη αξία. Επίσης στη Σουηδία υπήρξε η ίδια προσέγγιση γιατί δεν υπήρχε αυτή η αναπτυξιακή ε, πολιτική ε, οικοδόμηση συνεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προς το επόμενο βήμα, γιατί το 0,33% για τις νέες χώρες ή 0,7% για τις παλαιές χώρες δεν είναι πολλά χρήματα. Δεν είναι τόσο μεγάλος φόρτος όσο θεωρείται. Δεν έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στον προπολογισμό και χάνει κανείς την ε, τον πολιτικό του αντίκτυπο. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλάμε για 0,7 γιατί μιλάμε για την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών μας ε, πολιτικών. Θα πρέπει οι πολιτικές μας να είναι δυνατές, εύρωστες και να μην χάσουμε τη δυνατότητα μόχλευσης. Τώρα, ως προς μια πιο δεσμευτική πολιτική είναι πολύ πρόωρο να εικάσουμε, διότι ο προϋπολογισμός σχετίζεται με διαπραγματεύσεις και δεν θα ήθελα να εγγραφεί στον κοινοτικό νόμο το 0,7% τη στιγμή που δεν υπάρχει συνένεση. Αν υπήρχε συνένεση εντάξει, αλλά θα πρέπει να χτιστεί κάτι τέτοιο. Η Ιταλία είναι μια δύσκολη περίπτωση. Αλλά μέχρι το 2015 δεσμευτεί. Δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα και γι' αυτό θα ζητήσουμε τα, από τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν. Βεβαίως είναι ε, ένα χαμηλό ε, αριθμητικό στοιχείο, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε και με αυτό. Ως προς την Αιθιοπία, τις ελευθερίες και τη Realpolitik. Νομίζω ότι αυτό πάει πέρα από την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εμείς ήμασταν πολύ συνεπείς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ε, πρόκειτο για πρόβλημα με το Συμβούλιο. Οι δυσκολίες δεν σχετίζονται με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ούτε είναι η Realpolitik που φταίει γι' αυτό. Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Και πιστεύω ότι όταν διατυπώσουμε νέα στρατηγικά κείμενα θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, όλα αυτά είναι απόλυτα σαφή με βάση τη συνέργεια με τα κράτη-μέλη. Γιατί πάντα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και δεν μας το επιβάλλει αυτό η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά δεν υπήρξαμε πάντα συνεπείς. Γι' αυτό σας είπα ότι το όλο θέμα κινείται πέραν της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης, που τα κατάφερε πολύ καλά, υπέροχα θα μπορούσα να πω στην Αιθιοπία. Πρόκειται για μια εξελικτική πολιτική, το οποίο σημαίνει ότι όταν έχουμε χώρες όπως την Αιθιοπία θα πρέπει να συμφωνήσουμε και για έναν οδικό χάρτη και για θέματα που δεν μας έχουν ικανοποιήσει. Ως προς τις χώρες ΑΚΕ, διαφωνώ. Αυτή η συλλογιστική αναπτύχθηκε από τις ίδιες τις χώρες. Βεβαίως έχει σημασία η ιστορία, αναμφίβολα, αλλά οι ίδιες οι χώρες το πρόθεσαν. Και αν αρχίσουμε με καταργήσεις, αυτό σημαίνει ότι αυτό δημιουργεί σε παρανοήσεις. Είναι σαν να τους λέμε εμείς σας δημιουργήσουμε, εμείς σας καταργούμε. Ας αφήσουμε αυτό το σκεπτικό ακέ. Το ζήτημα είναι τι ρόλο παίζουν οι χώρες ε, ΑΚΕ πέρα από τον πολιτικό διάλογο, διότι προωθείται αυτός ο διάλογος. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί μπορούμε να δράσουμε αλλά ως προς την έννοια των χωρών και την θέλουν και θα το συζητήσω με τους ε, πρεσβευτές των χωρών και αύριο. Είναι δικό του σκεπτικό και δεν θα πρέπει να το καταργήσουμε γιατί εξαρτάται από αυτούς. Δηλαδή θα μπορούσαν, το, οι χώρες ΑΚΕ θα υπάρχουν ακόμα και αν δεν υπάρχει πια η Συμφωνία Κοτονού. Υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση ως προς αυτό το θέμα. Ως προς την αναθεώρηση γενικά, η συνένεση είναι πολύ καλή βάση και το 0,7% είναι ένα βασικό σημείο έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση και μεγαλύτερη δέσμευση. Θα δούμε πού θα οδηγήσει, αλλά νομίζω ότι το έγγραφο είναι εξαιρετικό, αλλά δεν είναι ε, πάντα εφικτό. Θα πιέσουμε για το 0,7 και για το Παγκόσμιο ε, Ταμείο έχουμε πολύ καλή συνεργασία, θα το δούμε οριζόντια και με θέματα και ως προς θέματα υγείας. Τώρα, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Η δική σας εποπτεία είναι ζωτική σημασία σαν σημείο κίνησης, διότι όταν επέλθουν συμφωνίες, έχει μεγάλη σημασία να είναι σωστό το σημείο εκκίνησης. Εάν είναι σωστό και εάν υποστηρίζεται και από την κοινωνία των πολιτών, θα στεφθεί από επιτυχία. Διαφορετικά δεν θα οδηγήσει σε ε, καλά αποτελέσματα η εξωτερική δράση θα πρέπει να είναι ένα σημείο αριστείας, δηλαδή δεν μεταφέρουμε ε, τους πόρους μας, απλώς επαναδημιουργούμε μια ευρωπαϊκή πολιτική με βάση την ποιότητα και την διαφάνεια. Και νομίζω ότι η Βαρόνη Άστον πιστεύει ακράδαντα ότι θα τα καταφέρει. Χρειάζεται χρόνος. Οπωσδήποτε χρειάζεται χρόνος, αλλά χρειαζόμαστε υποστήριξη εκινώντας από αυτό το, το σημείο. Ως προς το, το ερώτημα του κύριου Κάσμαν, φυσικά πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα. Όλα τα δικαιώματα είναι θεμελιώδη. Έχει σημασία πώς τα αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχουν πρωτογενή και δευτερογενή ανθρώπινα δικαιώματα κατανοούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αρχή αυτή και αυτό είναι το σημείο κίνησης. Πολλές φορές λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι από τη μία πλευρά η εξουσία από την άλλη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται η κοινωνία μας. Θα πρέπει να συμφωνούμε τι κάνουμε με την πολιτική Εάν ε, καταπολεμήσουμε αυτό το σχετισμό έχουμε αποτύχει. Εάν υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων σε μια χώρα, τότε θα πρέπει να αποσυρθούμε ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά για να συμφωνήσουμε θα πρέπει να υπάρχει πολιτικός διάλογος. Η Συμφωνία του Κότονου θα εστιάσει την προσοχή σε αυτά τα θέματα συζητήσεων. Πρόκειται για μία αμφίδρομη πορεία, διότι ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλη πορεία μπροστά μας. Θα πρέπει στην άλλη πλευρά να δώσουμε την ευκαιρία να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Άρα μπορούμε να το επιτύχουμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ως προς την θέση του Συμβουλίου, έχουμε ένα πολύ καλό προσχέδιο και αν συμφωνηθεί θα είναι αρκετά συνεπές και δυνατό. Άρα δεν αποσύρεται το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Ανάπτυξης έχει κοινά θέματα με το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών. Αλλά όλοι καταβάλουν σοβαρές ε, προσπάθειες. Έχουμε 40 χρόνια προϊστορία. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό το σκεπτικό. Για το θέμα της Προέδρου δεν το γνώρισα, λυπάμαι πάρα πολύ, θα το διερευνήσω. Ελπίζω να ε, αποστείλω Τέλονται εμπειρογνώμες. Κανένας δεν μπορεί να διώκεται για τη γνώμη του. Τιμώ οποιονδήποτε συνεργάζεται μαζί μου. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτή είναι η βάση της δημοκρατίας. Θα το συζητήσω σήμερα στο Διευθυντήριο. γιατί είναι επονίδιστο αυτό που συνέβη. Ως προς τις επενδύσεις στη Ζάμπια, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, θα το κοιτάξω. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία για να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις, διότι δεν θα γίνει δεν θα γίνει μεταφορά χρημάτων από, τις υπεράκτιες, από υπεράκτιες επιχειρήσεις. Αυτό οπωσδήποτε δεν πρέπει να γίνει. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο να τηρήσουμε και στενότερη συνεργασία μεταξύ της, ε, των αντιπροσώπιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε τους στόχους μας καλύτερα, για να δούμε πώς έχουν οι χρηματοδοτικές ροές. Και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και με την ΕΤΕ. Για να δούμε πώς θα κινηθούν και τα Ηνωμένα Έθνη με τη συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα. δεν ε, έχουμε ε, φτάσει σε πολύ μεγάλες νίκες, μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Για το ε, κέρας του ελεφαντοστού νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, διότι εμείς υποστηρίζουμε πάρα πολλά θέματα στη Σομαλία, υπάρχουν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Σομαλία, υπάρχει το θέμα και με την πειρατεία, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Αν υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάθε δίκη στοιχίζει εκατοντάδες χιλιάδες για θέματα πειρατείας και τα σχετικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να χρειαστεί χρόνος, αλλά και η κατάσταση τελευταία 20 ετία έχει επιδεινωθεί. θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε ορισμένα θέματα, γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται. Το ίδιο ισχύει και για το Αφγανιστάν. Οι Αμερικανοί είπαν ότι θα αποχωρήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, μπορούμε να προωθήσουμε την κατάσταση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δαπανίσαμε τόσα δις ευρώ. Δηλαδή μου λέτε ότι τα δαπανίσατε και τι άλλο. Και σας λέω τίποτα, απλώς τα δαπανίσαμε. Ίσως χρειαζόμαστε αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό ισχύει και για το ευαίσθητο αυτό περιβάλλον. γιατί έχουμε να κάνουμε με αυτές τις προκλήσεις, όπως σας είπα, για την αναπτυξιακή μας στρατηγική. γιατί και η κοινότητα θα πρέπει να κατανοήσει πώς έχει το θέμα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε τι μπορούμε να καλύψουμε και τι όχι. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους και θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο feedback. Και αυτό σημαίνει ότι θα ε, καλύψουμε ολόκληρο τον κύκλο του αναπτυξιακού προγράμματος. Σε αυτό το στάδιο για μένα έχει σημασία η αντίδρασή σας στο, στην επιστολή γιατί θα προωθήσουμε νέες σχέσεις και αυτό σημαίνει ότι θα κόψουμε τις γέφυρες εκεί όπου κινηθήκαμε διαφορετικά στο παρελθόν. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πού είναι οι προκλήσεις, ας πούμε στις αγροτικές περιοχές, στην Αφρική. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει τάση αστιφιλίας. Τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι πόλεις αν δεν δούμε θέματα, ας πούμε, ε, χωροταξικά, διότι όλοι θέλουν να ζουν όπως εμείς. Άρα υπάρχει μεγάλη ε, μετακίνηση προς τις μεγάλες πόλεις. Θα πρέπει να δούμε θέματα υγείας Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και αυτό το θέμα στο μέλλον. Η Αφρική αντιμετωπίζει τις ίδιες ε, προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ευρώπη 30, 40, 50 χρόνια πριν. Απλώς η κλίμακα είναι διαφορετική. Υπάρχει μία ε, εκρηκτική τάση ε, ανάπτυξης. Υπάρχουν δραστικοί ρυθμοί. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Έχουμε πάντα πολλούς εγγεγραμμένους. Θα ακολουθήσω δρακόντια μέτρα, 45 δευτερόλεπτα. Η κυρία Σνίμπερ Γιάστραμ. 45 δευτερόλεπτα και το τονίζω. Äh, äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Είπατε κάτι για τα μέτρα και την συνεργασία με άλλες χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας ή προσπαθειών συνεργασίας με Ινδία, με Κίνα, με άλλες χώρες δωρητές. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Merci beaucoup. Madame Ευχαριστούμε, questions, very quickly. Σύντομα. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει συνεκτική πολιτική. Ο ρόλο σα ε, ποιο είναι στην ε, ε, μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική και τη κοινή ελευτική πολιτική, τι θέλετε να πετύχετε στου τομεί αυτού και επίση η, η μεταρρύθμιση τη GSP που θα, προς τα που θα κινηθεί και τι ρόλο θα παίξετε. Είπατε για μια επιστολή που στείλετε, αλλά πώς μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε προς, την, προς μια πολιτική που θα βασίζεται και, στα, και σε ένα είδος δανεισμού παρά, και όχι μόνο στις ε, δωρές. Και επίσης πώς θα εξασφαλίσετε ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορέσει να μπει σε όλες τις ε, πτυχές της πολιτικής στα διάφορα νομικά κείμενα ε, και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στα στα δάνεια που δίνονται, στα, στους που δίνονται στις χώρες. Νομίζω ότι είναι τρομακτικό αυτό το ποσοστό που μας δίνεται τα 45 δευτερόλεπτα. Τι να πω σε 45 δευτερόλεπτα όταν διοργανώνονται τέτοιες ε, ε, ακροάσεις θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην ε, γίνεται μια τέτοια διοργάνωση, να μην υπάρχει αυτή η κακή διοργάνωση. Λοιπόν, ήδη είμαι στα 37 δευτερόλεπτα. Τι άλλο να πω μέχρι τα 45. Μιλήσατε για περιορισμούς της αναπτύξιακής πολιτικής. Καταρχήν, δεν ε, ξέρω κατά πόσο τηρούνται οι στόχοι της χιλιετίας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε μία δήλωση υποστήριξης προς, το Συμβούλιο κατά την επόμενη συναντησή του, έτσι ώστε να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους μέχρι το 2015. Επίσης, δεν υπάρχει επαρκής αλληλοσυσχετισμός βοήθειας ανθρωπιστικής και ε, οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή η ενδοκινοτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να βοηθήσει στην αναπτυξιακή αυτή πορεία. Δέχομαι αυτό τον κοινό προγραμματισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι μία εξωτερική ε, βοήθεια είναι, ε, α, δεν είναι πάντα αρκετή. Στην επόμενη συνάντηση με τις χώρες ΑΚΕ, λέει ο μιλητής και διακόπτη. Το δέχομαι. Το, το δέχομαι, το δέχομαι, εντάξει. Ε, δέχομαι αυτά που είπατε, αλλά θα πρέπει να δώσετε το λόγο σε άλλους. Ντέβα. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι σε 45 δευτερόλεπτα. Απλώς θα πρέπει να γίνει μια νέα συνάντηση έτσι ώστε να προωθήσουμε έναν καλός ε, διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή. Δεν, μπορώ να πω τίποτα σε 45 δευτερόλεπτα. Τι θέλετε τέλος πάντων. Yes, we will try to do that. And, um, uh, Madame Gre... Καλά, θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε άλλη συνάντηση. Κυρία Γκρές. Okay. Euh, monsieur le Commissaire, je, je vous remercie. Επίτροπε, δείχνετε εξαιρετική αποφασιστικότητα και ισχυρή θέληση να συνεργαστείτε μαζί μας και σας συγχαίρω. Όμως, άκουσα ότι όλα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των σχέσεων που υπακούν στους αναπτυξιακούς στόχους. Μιλάμε για την ενσωμάτωση των ηθαγενών ε, των γενών πληθυσμών, των γυναικών, με τις δράσεις μας θα μπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα στην παγκόσμια οικονομία μας, λέτε. Πολύ ωραία. Αλλά θα αναπτυχθούν και οι κρατικές υπηρεσίες, η πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, στην ε, επιστημιστική κυριαρχία. Πώς ακριβώς ε, θα εγγυηθείτε ότι οι πολιτικές μας θα είναι υποφελείς ε, για τους πολίτες. Και κάτι άλλο, ε, ας δούμε την επικαιρότητα, γιατί είναι σημαντική. Προτίθεστε να υιοθετήσετε μια πολιτική προαγωγή ενό κοινωνικού προτύπου, ενό αναπτυξιακού προτύπου που θα βασίζεται ε, στα ε, ατομικά δικαιώματα. Διακόπτει η Πρόεδρος. Η κυρία Κορτή, ευχαριστώ. Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας να γίνουν πιο ε, αποτελεσματικά να μην υπάρχει κατακαιρματισμός αναπτυξιακής βοήθειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στην ανάπτυξη των γενών κοινοτήτων και ερωτώ πώς ακριβώς θα έχουμε ε, πώς ακριβώς θα αξιοποιήσουμε τα κονδύλια που δαπανούμε σε κάθε χώρα πραγματικά. Ευχαριστούμε η κυρία Τόγια. Ε, ε Και εγώ θα μιλήσω για τον τρόπο ε, δαπάνησης των πόρων. Ξέρω ότι όλοι προσπαθούμε να φτάσουμε στους απότερους στόχους. Να φτάσουμε σε κάτι το σωστό. Στη, στη χώρα μου η κατάσταση είναι πολύ επώδυνη. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορείτε να κάνετε σαν Κομισιόν μεταξύ ε, του τι δεσμεύσεις αναλαμβάνουμε εδώ και τι κάνουν οι χώρες. Η καλή διακυβέρνηση σημαίνει ότι γίνεται και χρηστή χρήση ε, χρημάτων. Δεν θα πρέπει να κατασπαταλάμε το δημόσιο χρήμα τι συγκεκριμένες δεσμεύσεις ε, μπορείτε να αναλάβετε έτσι ώστε να μην γίνεται κακή δαπάνηση των πόρο. Ο κύριος Βένσον, τέλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να τονίσουμε ότι πέρα από τις θεμελιώδει ελευθερίες ε, υπάρχει το σημαντικό ποσοστό 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Εγώ νομίζω 1% πρέπει να είναι. Δεν χρειάζεται να με πέσουμε στο 0,7%. Όλοι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τα κόμματα στις χώρες τους. Εκεί πρέπει να ασκήσουν πίεση, όχι μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσουμε για να μείνουμε στο 1% ή να πέσουμε τελικά στο 0,7%. Ευχαριστώ, Επίτροπος. Θα απαντήσει. very, very short. Ναι, να απαντήσω σύντομα για την, ε, κυρία, για την ερώτηση της κυρίας Γιάστρομ με, την, ε, με τις ΕΠΑ έχουμε συγκεκριμένη πολιτική, ε, επιστημιστική βοήθεια, κλιματικές αλλαγές και ως το της χιλιετίας είναι τρεις στόχοι με τις ΕΠΑ. αλλά εμείς δεν θέλω να, δεν, έχω, δεν θέλω να δείχνουμε την εικόνα ότι εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε τα λεφτά και όλοι οι άλλοι κάνουν τη δουλειά. για την κυρία Κάλλας μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Βιωσιμότητα είναι η απάντηση. Για αυτό θέλω εγώ. Συνολική βιωσιμότητα και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, παγκόσμια βιωσιμότητα για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Όντως, αυτό που ρωτήσατε θα έπρεπε να εμπίπτει στον τομέα της ε, αναπτυξιακή βοήθειας. Και έχω συζητήσει αρκετά και με την συνάδελφο για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά το θέμα δεν είναι η... Ε, προσπαθούμε να έχουμε λίγο χωριστά τους προπολογισμού αυτά τα 2,4 δισεκατομμύρια, α πούμε, δεν θέλω να βγουν από ένα ταμείο και να πάνε σε ένα άλλο. Θα πρέπει να είναι κομμάτι της ε, κλιματικής αλλαγής. Αλλά τουλάχιστον ε, στην ε, αρχή ας, ξέρουμε ότι υπάρχουν επιπλέον χρήματα που θα έρθουν, ε, που θα προκύψουν. Πρέπει να είναι όντως mainstream η πολιτική, κεντρική πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Για την ενέργεια τώρα, θέλω να σας παρουσιάσω μέχρι το τέλος του χρόνου κάτι πιο συγκεκριμένο για τον κύριο Γκερέρο. Έχουμε το 0,7 στην ανακοίνωση και ελπίζω να το ενισχύσει, να το υποστηρίξει συγγνώμη, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Φυσικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για την συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε, την πιο εντελεχή. Το η επιστολή μου δίνει τη δυνατότητα σε, όλα τα κρατημέ... σε όλους τους ε, ευρωβουλευτές συγγνώμη, να δώσουν την άποψή τους και βεβαίως εγώ ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε ε, παρόλο που έχω πολλές ε, υποχρεώσεις, ταξιδεύω συχνά και εσείς επίσης ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια ημερομηνία και όποτε και είναι αυτή εγώ ευχαρίστω θα έρθω εδώ ακόμη και όλη τη μέρα αν θέλετε γιατί εντάξει προφανώς δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα θέματα μέσα σε 45 δευτερόλεπτα Αυτό που ρωτάει η κυρία Γκρέζα. Ε, ναι, φυσικά είναι ουσιώδες αυτό που ρωτάτε. Όταν πάμε στον τομέα τη ε, οικονομική ανάπτυξη, τη ε, δημιουργία θέσεων εργασία, δημιουργούμε νέου κινδύνου. Παίρνουμε λοιπόν ένα ρίσκο. Αλλά αν αφοσιωθούμε μόνο στα ε, φτωχά στρώματα της κοινωνίας δεν κάνουμε τίποτα. Το θέμα είναι να αλλάξει η γενικό νοοτροπία της κοινωνίας όλων των στρωμάτων. Αν θέλουμε να λύσουμε το θέμα της ε, ε, φτώχειας πρέπει να, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι το θέμα να δώσουμε λεφτά στους φτωχούς και τέρμα. Πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων η πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχουν χώρες που να μπορούν, στην Αφρική που να μπορούν να ε, αναπτυχθούν βιώσιμα. Η Νότιος Αφρική α, ε, κινείται, αναπτύσσεται αρκετά δυναμικά. Είναι μεγάλη λοιπόν η πρόκληση. Αλλά πρέπει να περάσουμε έτσι πολύ πόνο για να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ε, εκεί πρέπει να γίνει η συζήτηση. Τι κάνουμε, δίνουμε έτσι ένα έμβασμα εδώ, ένα έμβασμα εκεί για να βοηθήσουμε τώρα έτσι βραχυπρόθεσμα ή κάνουμε μια εκβάθρον αλλαγή για όλη την κοινωνία. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Η αλλαγή της κοινωνίας μπορεί να γίνει μόνο αν το δούμε το θέμα συνολικά. Τώρα, για το αντίκρισμα που έχουν τα χρήματα που δίνουμε. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία. Αν θέλουμε να επενδύσουμε κονδύλια Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα που περιμένουμε από αυτά τα κονδύλια και πρέπει να, να δείξουμε και στην κοινωνία ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα που θέλουμε. Γιατί δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, στην εκπαίδευση. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα στην εκπαίδευση, στην υγεία επίσης. Αλλά όταν πάμε στην ε, ενίσχυση του προπολογισμού σε συγκεκριμένα προγράμματα, μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Για με τα κράτη-μέλη τώρα. Οποιοδήποτε, οποιοδήποτε μείωση γίνεται, ε, εντάξει, προφανώς είναι βλαπτική, αλλά η ανάπτυξη είναι μία από τις υποχρεώσεις προς τον κόσμο που έχουμε. είναι πολύ δύσκολο να λύσουμε προβλήματα όπως ας πούμε αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Αν μπορούσαμε πριν από 20 χρόνια να έχουμε μπει στην καρδιά του προβλήματος, δεν θα είχαμε χρειαστεί να δαπανίσουμε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Τώρα είναι, έχουμε πολύ περισσότερες δυσκολίες και φυσικά όσο περνάνε τα χρόνια και δεν λύνεται το θέμα, Πάρα πολλά προβλήματα θα προκύπτουν. Στη Σομαλία 20 χρόνια, χρόνια είμαστε εκεί πόσα πόσα, τι έχουμε καταφέρει. Αν, αν δίναμε στον κάθε Σομαλό τα λεφτά που έχουμε δαπανίσει γενικώ για τα προγράμματα που έχουμε κάνει στη χώρα αυτή, όλοι οι Σομαλοί θα ήταν πλούσιοι σήμερα. Τώρα για το κατά πόσο δαπανούμε σωστά τα κονδύλια νομίζω ε, έχω απαντήσει, οπότε... Ε, όπως ε, θέλετε, όταν, ε, όποτε θέλετε, εγώ μπορώ να ξαναέρθω και να σας απαντήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Πίμπαλξ γιατί παρέμεινε μαζί μας περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο και θα ε, διοργανώσουμε τάχιστα μία νέα συνάντηση έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει άνετα να υποβάλει ερωτήσεις και να λάβει και απάντηση βέβαια. Θα εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη πολύ σύντομα. Nous allons maintenant aborder le point 5 de l'ordre. Σημείο 5 της Μέσης Διατάξεως, ε, αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αναθεώρηση της ε, Συμφωνίας του Κοτονού. Ε, εκ μέρου τη ε, Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου, ο κύριος Μαρτίν Γιάγκουε είναι ο σύμβουλο ΑΚΕ στην μόνιμη αντιπροσωπεία του Βασιλείου τη Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα. Χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε για να γίνει ανταλλαγή απόψεων για την αναθεωρημένη συμφωνία Κότονου Είστε επιφορτισμένος με αυτό το φάκελο στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ισπανίας και ειδικεύεστε στο θέμα αυτό. Γνωρίζετε ότι οι διαπραγματεύσεις για δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού ε, αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή μας. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ ε, καθώς και ο βασικός διαπραγματευτής Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέβαλαν τακτικά αναφορά για τις εξελίξεις ως προς τις διαπραγματεύσεις. Ε, τώρα καταλήξαν οι διαπραγματεύσεις σε μια συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει να υλοποιείται το, η διαπραγματευτική της ε, έντολη εξ ονόματος του Συμβουλίου, οπότε το Συμβουλίο θα αποφασίσει αν θα επικυρώσει τη Συμφωνία του Κοτονού και θα ε, συνεχίσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει στις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Η επίσημη υπογραφή της ε, αναθεωρημένης Συμφωνίας του Κοτονού έχει προβλεφθεί για τις 22 Ιουνίου ε, στο Μεικτό Συμβούλιο Υπουργών και Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Οπότε δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα με τον εκπρόσωπο της Προεδρίας, της Ισπανικής Προεδρίας, τον κύριο Μαρτίν Γιάνγκιού. Σας δίνουμε τον λόγο για πέντε λεπτά και μετά θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ. suis désolée, je n'étais pas consciente qu'elle n'était pas dans la salle. Donc, je souhaite la bien... Ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ότι είχατε ήδη μπει στην αίθουσα και τα είπα όλα αυτά. Τέλος πάντων, σας καλωσορίζω και σε... Σας δίνω ε, ε, απευθεία το λόγο για να μα μιλήσετε για πέντε λεπτά για τα τελευταία στάδια διαπραγματεύσεων για την αναθεωρημένη συμφωνία Κοτονού και να μας ενημερώσετε για τα τεκτενόμενα στο Συμβούλιο. Sí. Eh, muy buenos días, señora presidenta del Comité DEVE, señores. Κυρίες και κύριοι, Κύριοι ε, ε, Ευρωβουλευτέ, ονομάζομαι Μαρτίν Γιάγκουε και είμαι στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ισπανίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχολούμαι με θέματα ΑΚΕ. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ενώπιον σας τη σημερινή αυτή ημέρα για να σας εξηγήσω από πλευράς της Προεδρίας πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και ποια ήταν τα τελικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τις χώρες ΑΚΕ για την δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού και ποιες είναι οι προοπτικές που διανοίγονται μετά από την αναθεώρηση αυτή. Έχω πέντε λεπτά νομίζω για να σας εξηγήσω τη θέση της Προεδρίας και γι' αυτό εντάχει θα αναφερθώ στα θέματα τα οποία είναι πιο ενδιαφέροντα για εσάς και θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς τους Ευρωβουλευτές. Αυτή η δεύτερη αναθεώρηση του ε, Κοτονού άρχισε το 2009 και για 10 μήνες προβήκαμε σε μία ευρεία αναθεώρηση του, τύπου αλλά και τις ουσίες, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική διάσταση, τη θεσμική, την οικονομική και εμπορική, καθώς και την χρηματοοικονομική, χρηματοπιστωτική. Το τελευταίο ε, μέρος από την 1η Πρώτου του 2010 συνέπεσε με την Προεδρία και ασχοληθήκαμε πολύ περισσότερο με την Επιτροπή για να ασχοληθούμε με τα πλέον ουσιώδη ζητήματα μετά την αναθεώρηση του Κοτονού, μετά το τελικό κείμενο της 19ης Μαρτίου, έχουμε ένα πιο ε, εύρωστο κείμενο το οποίο βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την νέα αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα συνεργασίας και ανάπτυξης. Έχουμε μια ευρύτερη πλατφόρμα με βάση την κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Έχουμε εισαγάγει νέα στοιχεία που αποτελούν τμήμα των καθημερινών μας σχέσεων με τις χώρες ε, ΑΚΕ για να αντιμετωπίσουμε τους στόχους χιλιετίας, την καταπολέμηση του AIDS, τα αναπτυξιακά προγράμματα, την αλληλευτική πολιτική, θέματα ασφάλειας καθώς και τις αλλαγές στον προγραμματισμό για το στο Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Και αλλάξαμε ορισμένα θεσμικά ζητήματα, δηλαδή ενισχύσαμε το ρόλο των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων των χωρών ΑΚΕ καθώς και το ρόλο της συνέλευσης ίσης εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΚΕ, όπου ε, συμμετέχετε ενεργά. Για τον έλεγχο των μεμονωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης για τις χώρες ΑΚΕ, το, λεγόμενο, το λεγόμενο Country Strategy Paper, καθώς και την επαλήθευση και έλεγχο εφαρμογή συμφωνιών οικονομικής εταιρικής συνεργασίας. Υπάρχει ένα βασικό θέμα που σχετίζεται και με τον πολιτικό διάλογο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μετά από πρωτοβουλία της ίδιας της ε, Κομισιόν, αφού ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάποια συγκεκριμένη στιγμή της διαπραγμάτευσης προσπαθεί αφήσαμε να εισαγάγουμε μια ειδική ορολογία στο άρθρο 8 για να μην γίνονται διακρίσεις με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτό ήταν ένα αίτημα που είχε ζητηθεί εδώ και πολύ και καιρό και ο Γενικός Διευθυντής του, του τμήματος αυτού της Κομισιόν είχε έρθει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και μέχρι τις 19 Μαρτίου ε, γινόταν συνεχής μνήα σε αυτό το θέμα, δηλαδή η μη διάκριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού. Τελικώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν η συμπερίληψη αυτή και φτάσαμε σε μία ε, συμβιβαστική διατύπωση με βάση το άρθρο 2 της ε, Παγκόσμιας Δήλωσης ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπήρξε και μία μονομερής δήλωση, γιατί αυτό το άρθρο συνδέεται με αυτή τη συλλογιστική μη διάκριση, δηλαδή για λόγους σεξουαλικών προτιμήσεων. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν και κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η συμπερίληψη στο άρθρο αυτό θα μας βοηθούσε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά για να μην υπάρχουν διακρίσεις λόγω, ε, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Η κυβέρνηση του Μαλάουι έδωσε χάρη σε όσους είχαν καταδικαστεί επειδή είναι ομοφιλόφιλοι. Υπάρχει και το θέμα της μετανάστευσης και η ειλικρινά η Προεδρία θα πρέπει να διαπιστώσει ότι δεν είχαμε ένα επικερδές αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το άρθρο 13 για θέματα μετανάστευσης έτσι ώστε να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε στοιχεία όχι μόνο ως προς τη νόμιμη μετανάστευση αλλά και τις παράνομες μεταναστευτικές ε, ροές και να ε, ενισχύσουμε και το κεφάλαιο της επανεισδοχής. Αυτό το θέμα κατέληξε κάπως στις τελικές διαπραγματεύσεις και μπορούμε να εργαστούμε μέχρι την τελική επικύρηση. Μπορώ να σας πω ότι αυτή η αναθεωρημένη ε, έκδοση που ε, επικυρώθηκε και υπεγράφει από τον Επίτροπο ε, Πίμπαλξ θα επικυρωθεί και στη συνάντηση που θα γίνει στο Ουαγκαντούγκου τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ και με μεγάλη, μεγάλη μου χαρά να σας απαντήσω. Si, Monsieur Cashman, vous avez la parole. Ευχαριστώ κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας που ήρθε σήμερα να μας εξηγήσει τα όσα συμβαίνουν. Ε, δεν ήταν μόνο ανησυχία το Κοινοβουλίο να ε, συμπεριλάβουμε το σεξουαλικό προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις και αυτούς που ε, νοσούν από το AIDS. Ξέρετε, δεν είναι δική μας εφεύρεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Εμείς εκπροσωπούμε απλώς τους πολίτες ε, των εκλογικών μας περιφερειών. Για το άρθρο 8 αποτύχατε ικτρά και είναι χειρότερη κατάσταση για τους εξή λόγους. Ε, είπατε στο Μαλάουι ότι εδόθη χάρη στους ε, δύο ομοφιλοφίλους. Μα ε, λάθος τα λέτε. Εμείς είπαμε ότι δεν θα κάνουμε, δεν θα στείλουμε δήλωση και έτσι περάσαμε μήνυμα σε αυτά τα οπισθοδρομικά κράτη τη, τη ΑΚΕ, ο, ότι δηλαδή παίρνουμε στα σοβαρά, δεν παίρνουμε στα σοβαρά τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, φιλοφίλων και φιλομεταβατικών. Εγώ ε, είμαι ομοφιλόφιλος και θα ήθελα να σας πω ότι αν είχαμε διαπραγματευτεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, θρησκείες, το, το γενετήσιο προσανατολισμό, την εθνοτική προέλευση, δεν θα είχαμε αποτύχει. Θα, εμείς ε, και εσείς δεν θα είχαμε στείλει αυτό το φρικτό μήνυμα στις χώρες ΑΚΕ, δηλαδή επειδή κάποιοι ε, ανήκουν στη μειοψηφία, ε, ε, υφίστανται όλα αυτά, αυτό το μήνυμα περάσαμε. Αντίθετα, θα είχαμε πει στις χώρες ΑΚΕ ότι αν τελικά δεν καλύψετε και το γενετήσιο προσανατολισμό, τότε θα υποβάλουμε δήλωση. Όταν είπαν οι χώρες ΑΚΕ ότι επίσης θα υποβάλουν δήλωση. Τι κάναμε εμείς, υποχωρήσαμε. Δεν είχαμε το θάρρος να υπερασπιστούμε τις αξίες μας που είναι οικουμενικές αξίες. Στην Αφρική και μόνο, μό, τουλάχιστον 38 κράτη απαγορεύουν τις σεξουαλικές σχέσεις ε, ε, ιδίου φύλου και κάποιοι επιβάλλουν και τη θανατική ποινή. Γι' αυτό το λόγο το να επικυρώσουμε αυτή τη συμφωνία ισοδυναμεί με το να πετάξουμε στα σκουπίδια ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και να πούμε ότι άνθρωποι σαν και εμένα, έτσι, αν ζούσα εγώ εκεί, δεν θα έχουν τις ίδιες αξίες και τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς πολίτες. Και τι, η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων ε, ε, ε, που βλέπουμε στο άρθρο 8 λέτε εσείς ότι συνιστά πρόοδο, όχι. Υπήρχε με στη συμφωνία η οικουμενική ε, διακήρυξη των δικαιωμάτων και τώρα δεν υπάρχει πια. Ε, επιδεινώθηκε η κατάσταση και διατηρήσατε αυτήν την ανησυχητική φράση mutual concern, ε, αμοιβέ ανησυχίες. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να πούν ότι εμείς ανησυχούμε για αυτό, αλλά το άλλο μέρος δεν ανησυχεί ο Λί Μισελ, ο Κάρολ Ντεγκούχτο σε χώρε όπω το Μπουρούντι, το Μαλάου, την Κένια, την Ουγκάντα υπερασπίστηκαν ε, τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα και τελικά εσείς υποσκάψατε το φανταστικό αυτό έργο τους. Είμαι σίγουρος ότι το Κοινοβούλιο τελικά θα την επικυρώσει τη σύμφωνη, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ιεράρχηση των ατομικών δικαιωμάτων και τα δικά μου τα δικαιώματα θα παραγνωριστούν και θα παραμεληθούν σε αυτή την τόσο κρίσιμη ε, στιγμή. Και θέλω όμως να πείτε στην Προεδρία ε, ότι είμαι καταπληκτικός φίλος αλλά και καταπληκτικός εχθρός επίσης ε, και θα προσπαθήσω να αποτρέψω την επικύρωση της συμφωνίας συνεργαζόμενος με τα κράτη ΑΚΕ. Άλλο ε, η ροή των κονδυλίων προς αυτές τις χώρες, αλλά είναι επικίνδυνο να επικυρώσουμε τη συμφωνία γιατί το βασικό σημείο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και περνάμε το μήνυμα επικοινώνηση στη συμφωνία ότι δεν αξίζουν τα δικαιώματα των ε, ομοφιλοφίλων να τύχουν τι ίδιε υποστήριξει. Συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά είναι οι προσωπικέ μου πεπιθήσει και μιλώ για την πραγματικότητα ότι αν ε, ήταν δυνατή η σύλληψη αυτού του ανθρώπου και καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθριξη, ε, φανταστείτε θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε ανάμεσά μας και εφόσον δεν συμβαίνει σε εμά γιατί να συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Πρέπει το αναθεωρημένο σχέδιο να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Κανείς ε, δεν πρέπει να είναι περήφανος ε, επειδή έχει επιτύχει κάτι θυσιάζοντας όμως τα δικαιώματα κάποιων άλλων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς, έχω μία ερώτηση για την ασφάλεια και για την ανάπτυξη. Ε, αναφερθήκα σε αυτά τα ζητήματα στην εισαγωγική σας παρουσίαση. Θα ήθελα να μιλήσω όλος ιδιαίτερος ε, για ε, το θέμα των διευκολύνσεων για την ειρήνη που και τις αντίστοιχες διατάξεις στην ισχύουσα συμφωνία Κοτονού και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες ε, ΑΚΕ. Στο μέλλον θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ίδιο τύπο ε, και θα συμπεριληφθεί λοιπόν ε, θα, αντίστοιχη διάταξη στην, στο αναθεωρημένο σχέδιο της Συμφωνίας Κοτονού που τώρα διαπραγματεύεστε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντέβα, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Κάσμαν. Θυμάμαι όταν ε, πολεμούσαμε το Απαρτχάιντ ε, στη Νότια Αφρική, όταν ε, μεταχειριζόμαστε διαφορετικά κάποιους ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για τους ομοφιλοφίλους που το έχουν επιλέξει, το ε, κόμμα των συντηρητικών έχει αναλάβει δέσμευση για ισότιμη μεταχείριση όλων. Και ο ηγέτης μας, ο νέος πρωθυπουργός, το τόνισε και πάλι. Οπότε, ε, κύριε Προεδρεύοντα, δεν μου αφήνει τα άλλη επιλογή. Θα πρέπει να ζητήσω από την κυβέρνησή μου να μην χρηματοδοτήσει ε, τη νέα συμφωνία κοτώνων. Ε, ε, το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε και πάλι τον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας ε, για τρία λεπτά κατά νότα το όριο για να απαντήσει. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα με βάση την απόλυτη υπεποίθησή μου του τι εκπροσωπώ. Μιλήσατε για τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Προεδρία και η κυβέρνηση ε, κατήχε ηγετική θέση ήταν στην εμπροστοφυλακή υπέρ της ισότητας όλων των ανθρώπων παρά τις ε, σεξουαλικές τους διαφορές. Αυτή είναι μία απτή πραγματικότητα, είναι μία πραγματικότητα που γνώρισα και εγώ και προσπάθησα να, σας ε, το, να το μεταδώσω αυτό στις διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για την ε, Προεδρία αυτή και για κάθε προεδρία οι σεξουαλικές προτιμήσεις ε, είναι ένα θέμα ύψης της ε, σημασίας και κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Πολλοί ήσασταν παρόντες στη Λουάντα, στη συνέλευση ίσης εκπροσώπησης και είδατε την αντίδραση των ε, βουλευτών από την Αφρική γυναικών και ανδρών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να ε, δεχτούμε τι θέλει και η άλλη πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμαστε από το στόχο μας. Το γεγονός ότι κάποιος εισαγάγει πολιτικό διάλογο δεν σημαίνει ότι εν μία νυχτή αλλάζουν νομοθεσίες, ε, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κυρωτικές σε ορισμένα αφρικανικά κράτη ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό. Αλλά όπως είπε και ο Επίτροπος Πίμπαλξ, θα πρέπει να προωθήσουμε μία πολιτική για, έτσι ώστε να εισαγάγουμε αυτό το στοιχείο σε όλα τα μέτωπα πολιτικού διαλόγου στις χώρες ΑΚΕ και νομίζω ότι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε, η ιδιόγλωσσα που χρησιμοποιήθηκε στο άρθρο 8 μας το επιτρέπει αυτό. Αυτή, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση των πραγμάτων. Γιατί έχουμε να κάνουμε με θεμελιώδη, ουσιώδη ζητήματα για όλους. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία της Κομισιόν να ε, εισαγάγουμε αυτή την, την, γλώσσα μετά από την θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει όμως καμία παγκόσμια συμφωνία που να έχει υπογράψει μια χώρα ΑΚΕ όπου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει και ο όρος της μη διάκρισης ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Γιατί για εκείνο με συγχωρείτε, έχετε ε, ε, υπερβεί το χρόνο σας. Δίνω το λόγο στον κύριο Κάσμαν για μια τελευταία απάντηση. Κάσμαν. Δέχομαι την ειλικρίνεια, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όταν υπογράφουμε διεθνείς συμφωνίες, με τις χώρες ΑΚΕ η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί τους ζητούμε να, μας, να δεχτούν μια συμφωνία μαζί μας, άρα υποβιβάζουμε τις δικές μας αξίες. Εάν η παγκόσμια δήλωση είναι τόσο αποτελεσματική και αν υπήρχε στην αιτιολογική σκέψη, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη καταστολή. Η συζήτηση θα συνεχιστεί, θα προσπιστούμε αυτές τις αρχές όπως κάναμε και εμείς θα πρέπει να υπάρχει προοδευτική στάση και το ξέρουμε, ότι το, ε, το κατέδειξε αυτό η Ισπανία ως προς το, ε, το θέμα αυτό των ομοφιλοφίλων. Δεν σας κρίνω για αυτά που κάνατε στις άλλες χώρες, στη δική σας χώρα, αλλά για αυτά που κάνετε για τις άλλες χώρες και είναι λυπηρή η πρόταση της Προεδρίας. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder au vote. Donc, point. Oui, c'est ça. Donc, nous allons modifier l'ordre du jour légèrement pour tenir l'ordre. Θα αλλάξουμε την ε, ημερήσια διάταξη κάπως για να κρατήσουμε το ωράριο της ψηφοφορίας. Άρα αφήνουμε το, την ερώτηση προς την Επιτροπή προς το τέλος. Το τέλος η ερώτηση της Κομισιόν. D'accord. Donc, le vote est électronique. Il faut que vous... Ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ αναζητήσετε τις κάρτες σας, σας αφήνω λίγο χρόνο γι' αυτό. On va faire un essai de fonctionnement de, des appareils. Θα κάνουμε μία δοκιμή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Ça marche. Bon. D'accord. Donc, on vote sur la réduction de la pauvreté et la création. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 18. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επί της 18. rejeté. Ah, je, de, pas de rejeté. Ah oui, excusez-moi. Rejeté. Chez lisais 21 pour. Monsieur 4. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε, με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Δικαστικό. Δηλαδή, as many amendments as possible. Μπορούμε να ψηφίσουμε αν μπλοκ όσε περισσότερες γίνεται. Τροπολογίες. From uh, 19 until από την 19 μέχρι πιάν δηλαδή λέει η πρόεδρος. It was just a general remark. Γενική είναι η παρατήρηση. Donc 19. Only 19. Only 19. I'm sorry, but uh, I, okay. 19. 19. Αρχίζει ψυχοφορία. ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 21 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Donc, euh, Απορρίπτεται. 22. Αρχίζει η ψηφοφορία.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 Ζητά από όλες τις υποανάπτυξη χώρες να προσχωρήσουν στην ατζέντα για τις μειονότητες έτσι ώστε να είναι ικανοποιητική η κοινωνική προστασία και ένας πραγματικός κοινωνικός διάλογος ιδιαίτερα όταν προσφεύγουμε σε έργα που απαιτούν εντατικά αναπτυξιακό δυναμικό. Ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Le vote clos. Pérez. Εγκρίθηκε. Ensuite, en bloc, ah, en bloc de 23 à 24. C'est compliqué ça. Donc, euh, Προτιμώ να τις βλέπουμε κάθε μία ξεχωριστά, λέει η Πρόεδρος, γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Είμαστε στην 23, ρωτάει η Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 23. Ah, euh- Ψηφίζουμε από την 20 μέχρι την 24. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Μετά ψηφίζουμε μέχρι πού, ρωτάει η πρόεδρος. Α, μόνο την 25. 25 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Donc, restez. Απορρίφθηκε. Nous allons voter l'amendement 26, 27. 26, 27 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Tout le monde a voté. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Donc l'amendement aura... Προφορική υπαρχμών 2. Μίτσελ. Μπορείτε να μας τη διαβάσετε, αν έχετε την καλοσύνη. D'accord. Ίσως οδηγεί σε σύγχυση. Είναι του κυρίου Μισελ, λέει ο κύριος Γκέρενς. Επειδή μιλάμε για σωστή διακυβέρνηση, ένα κράτος θα πρέπει να αγκιάται τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εκπαίδευση και στη δημόσια δίκηση, έτσι ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Adapté. Ensuite... Euh, Εγκρίθηκε. Ίσως μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις 28, 29 και 5. Τις 3, 28, 29 και 5. Όχι. Καλά, καλά, με συγχωρείτε. Υπάρχει διαφωνία. Άρα, 28. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ανταπτή. Εγκρίθηκε. Euh, Από την 5 μέχρι τη 14. Ωραία. Αρχίζουμε, τις ψηφίζουμε μαζί. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκαν. 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Tout le monde a voté. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 32. 32. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 25. Αρχίζει η ψηφοφορία. Tout Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Adapté. Εγκρίθηκε. Από την 29 ψηφίζουμε μέχρι την 38. Άμε συγχωρείτε, μέχρι την 36. 29 έως 36. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Adapté. Εγκρίθηκαν. 37. Πρώτο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Restez, moi je vois 12, ah oui, 12, Απορρίφθηκε. 38. Mm, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Από 40, 41, 42 συμφωνείτε μπλοκ. Ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2. On vote le compromis 2 jusqu'à 46. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vote en bloc jusqu'à 46? Συμφωνείτε από το Συμβασμό 2 μέχρι και την 45 και την 45. Συμφωνείτε? Ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Emploi 10. Ah, emploi 3. 10 emploi. 10 από emploi. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Donc 49. 49. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Rejeté. Απορρίφθηκε. 50. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ανταπτή. Εγκρίθηκε. 51. Ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Προφορική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. Πενήντα τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Προφορική τροπολογία 4. Κύριε Γκέρνα, θα μας τη διαβάσετε. Ζητά ουσιαστική επιπρόσθετη χρηματοδότηση ε, για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και της οικονομικής κρίσης σε αναπτυσσόμενες χώρες. <clears throat> Tout voté, le Ψήφισαν όλοι πέρα. Δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρα. Εγκρίνεται. 20 ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 της Επιτροπής Απασχόλησης και 26 ομάδων. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Συμβαστική 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Την 57 λέει η πρόεδρος. Εγκρίνεται η 57. Συμβαστική 6 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Από την 59 μέχρι την 63 ομάδων συμφωνείτε. Όχι, καλά, εντάξει από την 59 μέχρι τη 16 Επιτροπής Απασχόλησης τότε από κοινού. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνονται. 27. Ψήφιστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 17 της Επιτροπής Απασχόλησης. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Από πού μέχρι που θέλετε να τις ψηφίσουμε μαζί. Από την, 20, την 28 και την 60 μόνο. Ωραία, ψηφίστε. Πέρας. εγκρίνονται. Οι πέντε τώρα. Πρέπει να τη διαβάσετε. Προφορική τροπολογία 5. Α, δεν γίνεται. Δώδεκα της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, από την 61 μέχρι και την 63 μαζί, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. 64. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 65 καταπίτη. 13 της Επιτροπής Απασχόλησης, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6. Κύριε Γκέρνς, θα μας τη διαβάσετε από τον κύριο Λουί Υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια ε, ρεσιμότητα εφαρμόζονται και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη αλλά και για τα μέσα χρηματοδότησης ε, της αναπτυξιακής ε, βοήθεια. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική 7. Ε, α, 7 και 8. Α, 7, δεν μπορούμε να τις δούμε μαζί. Η 7. Ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε να τηρηθεί η πολλαπλή συμμόρφωση όπως προβλέπεται από την Συμφωνία Κοτονού. Ευχαριστούμε. Ε, μπορώ να τη δεχτώ αυτή την τροπολογία μόνο ως προσθήκη, όχι σε αντικατάσταση της προηγούμενης. Δεν σας άκουσα, θα το ξαναπείτε. Μόνο ως προσθήκη στο πρωτότυπο μπορώ να δεχτώ αυτή την τροπολογία και όχι σε αντικατάσταση.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 Προφορική τροπολογία 8. Διαβάστε τι μας σας παρακαλούμε κύριε Γκέρενς. Στα αγγλικά είναι. Δέχεται τη χρήση τη στήριξη μέσω του προπολογισμού. Όχι, κάνω λάθο. Τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και τα χρηματοδοτικά μέσα. Μα σα τη διάβασα, Πρόεδρε, ήδη την 8. Όχι, όχι, εγώ κάνω λάθο, λέει ο Τονίζει ότι και το ΕΤΑ και το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία για την ανάπτυξη πρέπει να πληρούν τα ίδια ε, κριτήρια εφαρμογή και πολλαπλή συμμόρφωση. Ευχαριστούμε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 68. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Αταπτή. Εγκρίνεται. 22 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. ομαδών από την 69 μέχρι και την 72. Θέλετε, όχι, μέχρι πού τότε. Όχι, ωραία, χωριστά, 69. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 70. Πέρας. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Ε, συγγνώμη, ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 74 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες. Εγκρίνεται. 75. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, 76 παρακαλώ. Πέρας. Να απορρίπτεται. 77. Ψήφιστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 79 μέχρι την 82. Μέχρι την 82 λέει η Πρόεδρος, τώρα διορθών λέει μέχρι την 81. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρα. Εγκρίνονται. 82 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 86 τώρα, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 87, άρχεται ψηφοφορία. Θέλετε να προσπαθήσουμε ομάδο να ψηφίσουμε από την 87 ως την 90. Όχι. Okay. 87 λοιπόν μόνη της ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Την 88 και την 89 μαζί, όχι. Καλά, 88 τότε. Πέρας. Εγκρίνεται. 89. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αν θέλετε την 91 και την 92 να τις ψηφίσουμε μαζί, όχι, καλά, 91. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 92. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 93. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 94. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 95 πέρας απορρίπτεται 96 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Πάμε στα recitals, στα ραπέντε. Πέρας. Απορρίπτεται. Έξι, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. τις αιτιολογικές σκέψεις 7, 8, 9 δεν μπορούμε όλες μαζί να τις ψηφίσουμε. Όχι, μόνο την 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 8 και 9 είναι ταυτόσιμες. Μαζί. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας απορρίπτονται. Προφορική τροπολογία 10. Κύριε Γκέρενς, θα μας τη διαβάσετε. Υποστηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ε, βούλησή τους να ε, έχουν τη μέγιστη δυνατή προσθέμενη αξία αυτό συνεπάγεται μια αναπτυξιακή βιομηχανική πολιτική, η οποία όμως πρέπει να υπάγεται στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στην προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε, ψηφίστε. Πέρας. Λοιπόν, Τροπολογία 10 για την αιτιολογική F. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 13, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 11. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Ένα και δύο μαζί τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνατε. Θα ψηφίσουμε τώρα για την έκθεση, την τροποποιημένη έκθεση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Donc, euh, <coughs> un grand merci à Madame Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Θεοχάρου. Εργαστήκατε με εξαιρετικό τρόπο. Madam Πρόεδρε, μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδών για την ε, ε, ε, επόμενη έκθεση. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Είναι η έκθεση του κυρίου Μίτσελ. Ομαδών όλες οι τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πρέπει να ψηφίσουμε και τη γνωμοδότηση, τροποποιημένη γνωμοδότηση. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τώρα για την ε, έκθεση ε, του κυρίου Μίτσελ, ε, πάλι ομάδων της τροπολογίας, έρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Α, ναι, και για το τελικό σχέδιο πρέπει να ψηφίσουμε, όπως τροποποιήθηκε, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι, ωραία πέρας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Τέλεια, σας ευχαριστούμε κύριε Γκίμιτσελ για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε. Oui, on a le bon, bon nom de, de la personne. Hein? D'accord. Comme vous le savez, la Commission Développement. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας απέστειλε μία αντιπροσωπεία, κοινή αντιπροσωπεία, μαζί με την ΑΦΕΤ και τους προϋπολογισμούς στην Παλαιστίνη και στην ε, Γάζα την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, εκπροσωπηθήκαμε από τους Στρίφελ, Βέγγελ και την υποφαινόμενη. Μεταβήκαμε στη Γάζα και κατά την προσεχή μας συνεδρίαση θα σας ε, υποβάλουμε μία πλήρη εισήγηση Μπορώ να σας πω τι είδαμε βέβαια. Στην ε, Ιερουσαλήμ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την ε, κατασκευή του τείχους, βλέπουμε πώς δημιουργούνται αυτά τα προσκόμματα μεταξύ των πολιτών, δηλαδή ε, μεταξύ ε, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας. Η, το Ισραήλ αρνήθηκε, αρνήθηκε να περάσουμε από τα Αιγυπτιακά σύνορα και μπήκαμε στη Λωρίδα από τα σύνορα της Αιγύπτου, λέει η πρόεδρος. Χρειαστήκαμε 7 ώρες με το λεωφορείο για να το κάνουμε αυτό και επισκεφτήκαμε διάφορα μέρη, ήρθαμε σε επαφή με τους εκπροσώπους των τραπεζών της Παλαιστίνης. Δεν είναι δυνατόν να γίνει εμπόριο, νόμιμο εμπόριο, όλα έχουν παγώσει. Μόνο μέσω αγωγών μπορεί να γίνει, μέσω τούνελ μπορεί να γίνεται το εμπόριο. Και τα ε, κτίρια που κατασκευάζονται υπό την ε, γίδα της Σούμρατ έχουν σταματήσει εδώ και δύο χρόνια. Δεν υπάρχει τσιμέντο. 1.200 κατοικίες έχουν σταματήσει να κατασκευάζονται. Ζουν λοιπόν σε επισφαλείς καταβλισμούς οι κάτοικοι και Εκεί διαμένουν 10.000 άτομα γιατί τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να αγοράσουν τσιμέντο από την μαύρη αγορά. Επίσης στη ε, Γάζα οι κατασκευές γίνονται με τσιμέντο που έχει αγοραστεί παράνομα. Ήρθαμε σε επαφή με τους εκπροσώπους ε, της UNRAD που μας ε, μίλησαν για τις δυσκολίες της καθημερινής επιβίωσης και δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε ε, Είχαν Είχαμε έξι ναυτικά μίλια για την αλία. Οι ε, σαρδέλες δεν ε, περνάνε, όπως ξέρετε, στις παράκτιες περιοχές. Αλλιεύονται στα τρία μίλια και πάνω. Αλλά τώρα οι Ισραηλινοί τους απαγορεύουν να αλλιεύουν εκεί. Υπάρχει μεγάλη διατροφική κρίση. Το 80% του πληθυσμού ε, διαβεί από τη βοήθεια της UNRAD. Σήμερα καλέσαμε την κυρία Βιρζίνια Βιλάρ που εργάζεται εδώ στα γραφεία της Ούμουρα στις Βρυξέλλες για να μας μιλήσει για την ανθρωπιστική ε, κατάσταση και βοήθεια στη λωρίδα της ε, Γάζας. Η πλήρης ε, αντιπροσωπεία ήδη από την Παρασκευή έχει συντάξει ένα ανακοινωθέν τύπου για να ζητήσει την άρση του αποκλεισμού στη λωρίδα της Γάζας, διότι είναι αντιπαραγωγικός αυτός ο αποκλεισμός ε, υποβοηθά τη μαύρη αγορά και καταστέλει τα δικαιώματα του πληθυσμού που απαρτίζεται κατά 50% από παιδιά κάτω των 18 ετών. Συναντήσαμε εξαιρετικούς ανθρώπους που προσπαθούν να καταστήλουν τη βία στα σχολεία υπό δύσκολες συνθήκες. Κάθε χρόνο προσέρχονται 6.000 παιδιά στα σχολεία, αλλά λόγω αποκλεισμού δεν μπορούν να αμυφθούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, γι' αυτό ζητήθηκαν περισσότερα κονδύλια. Με, αυτή την, με αυτό το ανακοινωθέν τύπου ε, ομόφωνα ζητήσαμε την άρση του αποκλεισμού και μάθαμε επιστρέφοντας στη Γαλλία και στις άλλες χώρες. Μάθαμε για την επίθεση του Ισραηλινού στρατού των ενόπλων δυνάμεων κατά της νιοπομπής, η οποία μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για να καταπραίνει το... την επώδυνη αυτή κατάσταση και ζητήσαμε να διενεργηθεί μία ανεξάρτητη διεθνής έρευνα για να δούμε πώς έλαβαν χώρα τα γεγονότα. Το Ισραήλ κατέκλυσε τα ΜΜΕ Γι' αυτό δεν έχουμε αντικειμενική θεώρηση του τι συνέβη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνήλθε χτες και πρότεινε μία αντικειμενική διεθνή έρευνα, αλλά δεν την επέβαλε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η μετάβασή μας ήταν ε, πολύ μεγάλη σημασίας. Υπήρξε μεγάλη αναγνώριση από τον ε, εγχώριο πληθυσμό της παρουσίας μας. Σας προτείνω σε μία επόμενη συνάντησή μας να ε, ζητήσουμε τη συνάντηση με τον υπεύθυνο της ΟΥΡΑ για να μας μιλήσει για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, τον κύριο Τζον Κίνγκ. Έχει μεγάλη σημασία για τα ποσά που δαπανάμε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήταν πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Η κυρία Βιλάρ όμως έχει πληροφορίες από τη Γάζα. Σας δίνω το λόγο για 5 με 10 λεπτά. Um, Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζολή. Ευχαριστώ που καλάσατε την όνορα στην σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τα μέλη της αντιπροσωπείας που επισκέφτηκαν για την επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα και την υποστήριξη στη δουλειά μας. Ξέρω ότι τα περισσότερα μέλη γνωρίζουν ε, την ε, εντολή της ΟΝΡΑ και για την παροχή υπηρεσιών για 4,7 εκατομμύρια προσφύγων στην περιοχή. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, θα πάω κατευθείαν στις ε, πληροφορίες για την ανθρωπιστική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Για να σας το δείξω αυτό, αφήστε, να, αφήστε με να σας πω κάποια στατιστικά στοιχεία. Από το 1,5 εκατομμύριο ε, άτομα που διαμένουν στη Γάσα, σε μια, σε μια έκταση 40 10 χιλιόμετρα, 80% πρέπει να ενισχυθούν με κάποια είδους βοήθεια. Το, σχεδόν όλο το ποσοστό αυτό είναι ανέργη στα σημεία ε, διέλευσης περίπου 19% των ε, επιχειρήσεων, 90% των επιχειρήσεων έκλεισαν, 94% των εργαζομένων έχασαν τη δουλειά τους. 56% του πληθυσμού στη Γάζα είναι κάτω των 18 ετών. Τα σχολεία στη Γάζα έχουν περίπου χίλιους μαθητές, 50 μαθητές ανατάξει και κάποιες ακόμη πληροφορίες για την πρόσβαση. Οι ανάγκες αυτού του 1,5 εκατομμυρίου ατόμων πρέπει να καλυφθούν από 80 περίπου ε, φορτηγά την ημέρα. Οπότε σκεφτείτε από μόνοι σας ε, κατά πόσο είναι επαρκές αυτό ή όχι. Σε σύγκριση, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εκτιμήσει ότι τουλάχιστον 500 φορτηγά πρέπει να μπαίνουν στη Γάζα κάθε μέρα για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των Παλαιστινίων. Επίσης, περίπου 400 ε, φορτηγά των, μπήκανε στο, έμπαιναν κάθε μέρα στην Γάζα τον Μάη του 2007 πριν αναλάβει η Χαμάς και περίπου ε, τα διπλάσια έμπαιναν τον, ε, το 2005. Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις τα, για τα κατασκευαστικά υλικά, ε, μπογιές και τα λοιπά που χρειάζονται μετά τις ε, σειράξεις για την ε, αναδόμηση είναι πάρα πολύ περιοριστική, ίσως και απαγορευμένη η εισοδός τους. Αλλά ακόμη και πλαστικά παιχνίδια, σοκολάτες, ξύλα για έπιπλα, χυμή, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στη Γάζα. Θα διαβάσατε ίσως ότι σε μια, σε μια υποβολή εκθέσεως στο δικαστήριο περιλήφθηκαν, ε, προϊό... Ε, περιλήφθηκαν ε, έγγραφα που, που αναφέρουν την απαγόρευση, καθώς επίσης και ότι δεν καλύπτονται οι ελάχιστες θερμιδικές ανάγκες των πολιτών της Γάζας. Βέβαια το έγγραφο αυτό έχει παραμείνει εκρεμές και προς το παρόν μόνο 81 προϊόντα επιτρέπεται να εισέρχονται στη Γάζα, να μπαίνουν στη Γάζα. Δεν υπάρχει ε, πετρέλαιο ούτε διζελ για τα αυτοκίνητα από το 2008. Η μόνη πηγή ε, παροχής ενέργειας λαμβάνει μόνο ένα τρίτο ε, καυσίμων για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Ε, αέριο για μαγείρεμα δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο για να καλύψει το 50% των αναγκών γενική πρόσβαση σε καύσιμα επίσης πολύ περιορισμένη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει, υπάρχει μεγάλη ε, έλλειψη και υπάρχουν και, πολλές, ε, και πολλά blackout. Αυτό βεβαίω δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινή ζωή. Έχει επιπτώσει και στη δημόσια υγεία. Αν λάβετε υπόψη ε, την έλλειψη αυτού του, της συντήρησης του ηλεκτρικού, ε, των ανταλλακτικών. Ε, καταλαβαίνετε ότι το σύστημα, σύστημα υδροδότησης πάσχει, το ηλεκτρικό πάσχει και αυτό φυσικά έχει τεράστιες συνέπειες στη δημόσια υγεία. Επίσης, ε, επειδή ακριβώς οι απειλές είναι μεγαλύτερες, το σύστημα υγείας δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ επιτρέπει κάποια φορτηγά να περνούν, αλλά βασικές ανάγκες, βασικές, ε, βασικά προϊόντα για την υγεία δεν ε, επιτρέπεται να περάσουν. Δηλαδή πέρα από τα φάρμακα χρειάζονται εξοπλισμός, χρειάζονται ανταλλακτικά, χρειάζονται όλα αυτά, χρειάζονται συντήρηση. Και όπω είπα, χρειάζονται ε, υπηρεσίε εξυγίανση, χρειάζονται γιατροί που πρέπει να πάνε να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν για τη δουλειά τους. Χρειάζονται όλα αυτά ώστε το σύστημα να είναι λειτουργικό. Τώρα, για τα τούνελ. Λόγω του οικονομικού ε, μπλοκ που υπάρχει, είναι, τα τούνελ είναι η ε, γραμμή ζωής. Υπάρχουν περίπου 2.200 ε, τούνελ, γιατί έχουν κλείσει πάρα πολλά σημεία διέλευσης τα προϊόντα που μπαίνουν είναι σε πάρα πολύ ψηλέ τιμές που σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα αποκτήσουν οι πιο φτωχοί και πέρσι όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν για το φαγητό τους, για την οικογένειά τους και για τους ίδιους από 100.000 έφτασαν τους 300.000. Αυτό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θα θεωρεί το απαράδεκτο. Ο έχει δείξει με διάφορα πολιτικά προγράμματα ότι έχει το μηχανισμό για να μετρήσει τους, ε, τα θύματα αυτών, των, αυτής της κατάστασης. Η Ισπανική Προεδρία επανέλαβε χτες σε μια, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι θα βοηθήσει να ε, ενισχυθεί ε, η Γάζα μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Η κυρία Ζολή το είπε και πιο πριν και το είδαν και επί τόπου, ε, το εμπάργκο που έχει μπει στη Γάζα από το 2007 έχει δυσχεράνει ε, την κατάσταση για τους ε, Παλαιστινίου έχει αυξήσει τη φτώχεια, έχει αυξήσει την ανασφάλεια, έχει αποτρέψει την επανα, επαναδιάρθρωση του, την ανοικοδόμηση, έχει καταστρέψει το βιό των ανθρώπων, την οικονομική δραστηριότητα, η, το άνοιγμα των επίσημων συνόρων τη γάζα για να υπάρχει καλύτερη εισρωή ατόμων από και προ τη Γάζα και προϊόντων είναι ο μόνο τρόπο για να σταματήσει αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή. Το άνοιγμα λοιπόν των επίσημων συνόρων τη γάζα θα επιτρέψει να αποφευθούν και άλλε ε, κατα καταστάσεις όπως οι καταστροφές όπως η Αυτή είναι η θέση λοιπόν της ε, UNRWA για τις ε, ε, πράξεις βίας που είχαν, που υπέστησαν όσοι μεταφέρουν προϊόντα στη Γάζα. Ο Φιλίππο Γκράντε, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΝΡΑ, έχει αναφέρει ότι τέτοιες τραγωδίες, τραγωδίες μπορούν να αποφευθούν εάν το Ισραήλ ε, σταματήσει την αντιπαραγωγική ε, το, ε, το αντιπαραγωγικό μπλοκάρισμα της, της Γάζας, το εμπαργό το οποίο το ζητά όλη η διεθνής κοινότητα. Και επίσης υποστηρίζουμε την, την υποστήριξη του Συμβουλίου για την έρευνα που θα βασίζεται στα διεθνή πρότυπα. Έχει να κάνει αυτό και με, την, με το άνοιγμα των σημείων διέλευσης ε, που υπάρχει και δυνάμει του 18-16 ψηφίσματος του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσελ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την αντιπροσωπεία που μετέβει στη Γάζα και ευχαριστούμε το, την εκπρόσωπο της Ουνδραντ. Συμπονούμε, συμπάσχουμε με αυτούς που υποφέρουν. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά αυτό δεν γεμίζει την κοιλιά τους, ούτε δίνει φάρμακα στα νοσοκομεία. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ξέρουμε όλοι ποια θα είναι η έκβαση. Δύο κράτη, μία λύση με δύο κράτη. Δεν γίνεται αλλιώ. Για 30 χρόνια στην Ιρλανδία το ξέραμε ότι θα γίνει έτσι, αλλά τελικά ε, επειδή είμαστε και λίγο αργόστροφοι, κάποιοι εν πάση περιπτώσει, χρειάστηκαν 30 χρόνια για να καταλήξουν σε αυτή την ε, λύση. Από τη δική μου εμπειρία, πάντως ξέρω ότι οι έξωθεν ε, συστάσεις και επιταγές δεν συνιστούν προς θέμενη αξία και δεν φέρνουν καμία λύση. Αυτά θα ήθελα να τα πω εν είδη εισαγωγής. Είδα στην τηλεόραση την υπερβολική βία, σαφώς πέθαναν πολλοί άνθρωποι στα χέρια των Ισραηλινών στρατιωτών. Είδα βέβαια ότι τραυματίστηκαν ε, και αυτοί, ε, δηλαδή κάθονταν στην ουρά όλοι με όπλα για να τους βαρέσουν. Το είδα αυτό στα κλιπάκια. Και δεν είχαν μόνο αυτοσχέδια όπλα. Αυτό είναι σίγουρο. Πρόεδρε, όπως και εσείς, πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να γίνει ανεξάρτητη διεθνής έρευνα για το τι έγινε. Δεν μπορούμε ε, επιτόπου να τους αφήσουμε να μας σερβίρουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων. Αυτό είναι προπαγάνδα. Εμείς πρέπει να ερευνήσουμε, να βρούμε την αλήθεια. Αυτή πρέπει να μας απασχολεί. Δεν νομίζω ότι είναι τρόπος ε, ε, παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας αυτός, παρά τις καλές προθέσεις 250.000 ετών ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν βρεθεί στην έρημο γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στη Γάζα. Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Ε, τη χρειάζονται τη βοήθεια εκεί, τα παιδιά, οι άμαχοι. Πρέπει να ζητήσουμε από το Ισραήλ να ανοίξει τις πύλες. Ε, μπορεί βέβαια να αντιδράσουν θετικά ή όχι, ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οι Αιγύπτιοι πάλι άνοιξαν τα σύνορά τους ήδη. Ε, πρέπει έτσι να αρχίσουμε να τροφοδοτούμε με βοήθεια, δηλαδή πράγματα που χρειάζονται άμεσα, τροφή, φάρμακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος πρέπει να πούνε συλλογικά θα κινηθούμε τώρα, συλλογικά θα βοηθήσουμε. Επίση, Επίσης, ε, κάτι τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να μας πει τι έχει γίνει για αυτό το θέμα ενδοϊπηρεσιακά. Τι κάνει η Εκπρόσωπος, πώς δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ που εγγράψατε το σημείο στην ημερήσια διάταξη για τη Γάζα, γιατί είναι ιδιαίτερα ε, σοβαρή η κατάσταση. Είναι κρίσιμη η στιγμή. Έχουμε, μας έχει κολλήσει στον τοίχο η τελευταία εξέλιξη. Ε, ο ΙΕ, η κυρία Άστον, η αντιπροσωπεία ζήτησαν διεθνή έρευνα. Πρέπει να επομιστούμε τις ευθύνες μας. Χρήσιμη και η διπλωματία, αλλά δεν αρκεί αυτή η πίεση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί και συνεπώς δεν μπορούμε να προβάλλουμε μία συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να προβούμε σε δράσεις. 18 δις ευρώ ε, έχουν επενδυθεί από το 1995 μέχρι το 2007 για τις χώρες της Μεσογειακής ε, ε, Λεκάνης. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να προωθήσουμε στα πλαίσια της Euromed. Αλλά θα ήθελα επίσημα να ζητήσω εδώ η Επιτροπή Ανάπτυξης να ζητήσει από την Κομισιόν και το Συμβούλιο το πάγωμα της συνεργασίας με το Ισραήλ ε, επικαλούμενη τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλές ε, συμφωνίες εταιρικής οικονομικής συνεργασίας. Η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για την αποστολή μας. Θα πρέπει φυσικά να συνεχίσουμε να καθιστούμε σαφές ότι είναι πολύ κακή προσέγγιση, προσέγγιση του αποκλεισμού και στην Ιερουσαλήμ πήγαμε στη Χευρόν, στην Απλούς, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μας συνάντησε και ο Πρωθυπουργός Φαγιάτ. Είδαμε τι έκανε για τον ε, πληθυσμό και προσπάθησε να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να έχει περισσότερη επιρροή στον Παλαιστινιακό λαό. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν την ε, πολιτική Φαγιάντ. Επίσης είχαμε πολύ καλές ε, συζητήσεις με τον εκπρόσωπο της Σούναρα και θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι για την ανάπτυξη. Εμείς επιδοτούμε όχι μόνο τους Παλαιστινίους εντός και εκτός ε, κατεχομένων, γιατί μόνο πέρσι δώσαμε 500, ε, δόθηκαν συνολικά 500 δις. Εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές της Ούνρα έχουν 30% από το δικό μας προϋπολογισμό και οι άλλοι δωρητές, τα άλλα χρήματα προέρχονται από τις ΗΠΑ, από την Ορβηγία και λιγότερο από 1% από αραβικές χώρες. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να στήσουμε από την κυρία Άστον να βρει τρόπους για να πιέσει και άλλες αραβικές χώρες να συνεισφέρουν. Γιατί ο προϋπολογισμός είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να δώσουν 10.000 μισθούς για δασκάλους, γιατρούς κλπ. Αν δεν πάνε σε σχολεία της ΟΝΡΑ θα πάνε στα σχολεία της Χαμάς θα πρέπει να βρούμε τρόπο επιμερισμού αυτού του ε, βάρους. Και όλες και οι άλλες χώρες θα πρέπει να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ αρχής θα πω ότι η τωρινή κατάσταση είναι υπέρ των πλέον ανευθύνων, εκατέρωθεν. Δεύτερον, είναι απεχθής η κατάσταση εδώ και χρόνια, αλλά διαρκώς επιδεινώνονται. Τρίτον, θα ήθελα να εγκομιάσω την ούντρα για το, τα όσα έχει κάνει επιτόπου στη Γάζα. και να τονίσω ότι είναι αμερόληπτη η δράση της. Αυτό είναι κέριο χαρακτηριστικό της ανθρωπιστικής δράσης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεδομένων των αναγκών που μόλις εκθέσατε και των εμπορευμάτων που γίνεται να διακομιστούν, αυτός ο αμερόληπτος χαρακτήρας ακριβώς θα σας επιτρέψει να δράσετε επί τη βάση των αναγκών που ε, διαπιστώνεται επί τόπου, βλέπουμε ότι παραβιάζεται η αρχή της αμερόληπτης δράσης. Πρέπει λοιπόν να τηρηθούν οι βασικές αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει βέβαια η διάσταση της ασφάλειας, αλλά υπάρχει η ανθρωπιστική διάσταση και πρέπει να τις διακρίνουμε. Σωστά τα περί ασφαλείας. Και μπορούμε να πούμε ότι το τσιμέντο, παραδείγματος χάρη, η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς τάξεις για τους μαθητές, η πρόσβαση σε επαρκή ε, τροφή, δεν μπορεί να μην κατοχυρωθούν. Δηλαδή, επί της αρχής δεν μπορεί κανείς να αντιταχθεί στην ε, διακόμιση αυτών των βασικών αγαθών ε, στη Γάζα. Δεν, υπάρχει, δεν συντρέχει κανένας θεμητός λόγος για να διατηρείται η απαγόρευση που πλήττει τον πληθυσμό της Γάζας. Εγώ επισκέφθηκα τη Γάζα πριν από χρόνια και ήταν ήδη φρικτή η κατάσταση και σας είπα ότι διαρκώς επιδεινώνεται. Ε, στον πολιτικό μας διάλογο νομίζω ότι θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ του διαλόγου με, τους, με όσους έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά. Υπάρχουν και στις δύο εμπόλεμες πλευρές και σαφώς διακρίνονται από την πρώτη κατηγορία των ανευθύνων που ανέφερα στην αρχή της παρέμβασής μου. Η πρωταρχική μας αποστολή πάντως πρέπει να είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και συμφωνώ με την πρόταση του Γκέι Μίτσελ ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Αίγυπτο γιατί από εκεί υπάρχει πρόσβαση οπότε η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεργασία με την Αίγυπτο ούτω ώστε να υλοποιηθεί ε, η δεδηλωμένη μας αυτή πρόθεση. Ευχαριστούμε ο κύριος Κάσμον τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση, για την επίσκεψή σας, για την αποστολή. Συμφωνώ με αυτά που είπαν και τα υπόλοιπα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Όντω πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη έρευνα, πρέπει να γίνει. Και χωρίς το εμπάργο, η τελευταία αυτή ε, καταστροφή μπορεί να είχε, τραγωδία μπορεί να είχε αποφευχθεί. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε με τους μετριοπαθείς, αλλά συνήθως φέρνει αυτό αντίθετα αποτελέσματα, ε, φέρνει αντίδραση και αύξηση του εξτρεμισμού. Οπότε αυτή η πολιτική δεν λειτουργεί από ό,τι φαίνεται. Η μόνη στιγμή όπου το Κοινοβούλιο ε, ψήφισε να ανασταλεί η Συμφωνία Σύνδεσης ήταν η προηγούμενη συμφωνία σύνδεση με το Ισραήλ και νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε να φέρουμε ένα κείμενο εδώ στο Κοινοβούλιο με μια τέτοια σύσταση. Γιατί εκτός και ε, μόνο αν επιβάλλουμε κάτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα, μόνο τότε θα μπορέσουμε να γίνουμε πιστικοί για το πόσο σημαντικά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο συντονιστή από την ομάδα μα κάθεται εδώ στα αριστερά μου, οπότε φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουν και οι συντονιστέ αυτό. Αλλά πραγματικά είναι εξαιρετικά κρίσιμο το ότι ήσασταν εκεί και εξαιρετικά ευτυχέ ότι ήσασταν εκεί αυτή τη στιγμή ώστε να έχουμε μια εκ των έσω εικόνα και να δούμε πώ μπορούμε να απαντήσουμε. Η πραγματικότητα είναι όμω, όπω είπε και ο κύριο Μίτσελ, όταν βλέπω εγώ την Ιρλανδία, α πούμε, και το πώ δημιουργήθηκε το κράτο του Ισραήλ όλα προέκυψαν από, τις, ε, από διαπραγματεύσεις με ανθρώπους που δεν θα διαπραγματευόσουν ποτέ αν μπορούσες να το επιλέξεις. Κάποιοι ονομάζονται υπερασπιστές, μαχητές της ελευθερίας. Από όποια πλευρά και αν έρχονται όμως, τα επιχειρήματά τους πρέπει να απαντηθούν, γιατί αλλιώς η τραγωδία αυτή θα συνεχιστεί. Ναι, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο, ε, ο κύριος Γκέρενς και ο κύριος Κάσμαν. Ήθελα να τονίσω κάποια σημεία. Ε, η επιδρομή πριν από λίγες μέρες δεν πρέπει να συγχέεται με την κατάσταση στη Γάζα. Ε, δεν είναι η σχέση αιτίου αιτιατού. δηλαδή, η, ο αποκλεισμός δεν θέλουμε να αρθεί μόνο και μόνο λόγω της επιδρομής, θέλουμε να αρθεί επειδή ζουν σε ιδεχθείς συνθήκες ε, στη Γάζα. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση όσο υπάρχει ο αποκλεισμό. Οπότε, συμφωνώ με τον κύριο Γκέρεν, άλλο η ασφάλεια και άλλο η ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι θα σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα τη ανθρωπιστική ε, βοήθεια. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να προσθέσω μόνο. Η κυρία να ευχαριστήσω και εγώ όλους όσους συνέβαλαν με τις πληροφορίες τους και εμείς νομίζω ότι ως ε, μέλη της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης θα πρέπει όντως να κάνουμε τη δική μας, συναδόση δώσουμε τη δική μας συμβολή, να φτάσουμε σε ένα ψήφισμα για την αναθεώρηση ίσως της ε, Συμφωνίας Σύνθεσης με το Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό το αίτημα του ε, συναδέλφου Μίτσελ για την ε, ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα πρέπει να εξετάσει το τι γίνεται θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Ε, υπάρχουν διάφορες αναφορές βέβαια για το πώς προχωρούν, πώς έγινε η κατάσταση, πώς κατέλαβαν τα πλοία κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι Δεν θα, πρέπει να καταρχήν να δούμε τι έχει γίνει πραγματικά γιατί έχουν υπάρξει βίντεο στο ίντερνετ που μπορεί να είναι παραποιημένα, που μπορεί να είναι ψεύτικα. Που υπάρχουν ε, επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν υπάρξει άνθρωποι πληγωμένοι, άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Δεν μπορούμε έτσι απλώ να το προσπεράσουμε. Πρέπει να έχουμε τα αντικειμενικά γεγονότα. Εγώ πάντα λυπούμε γιατί είμαστε πάντα ανασφαλείς για το τι, πώς αξιολογούμε αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η πολιτική της, Ισραήλ, της, πολιτική, της κυβέρνησης του Ισραήλ δεν μπορεί να είναι ίδια με τον αντισημιτισμό. Το κράτος του Ισραήλ μάλλον στο, του Ισραήλ δεν ε, ζουν μόνο Εβραίοι, ζουν και άλλοι. Οπότε λοιπόν πρέπει να δώσουμε πηγόντως ένα μήνυμα προς τον πληθυσμό του ε, Ισραήλ, προς τους ανθρώπους που είναι μετριοπαθείς, που ζουν στο Ισραήλ και θέλουν αλλαγή της ε, κυβέρνησης και θέλουν αλλαγή της πολιτικής. Πρέπει λοιπόν και εμείς να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή, η, αυτό το αίτημα για την υποστήριξη των, ε, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχύει και από τις δυο μεριές. ώστε να δούμε γιατί έχει ο πληθυσμό του Ισραήλ αυτή την αμυντική στάση πάντα. Εγώ είμαι από μια χώρα η οποία είχε χρόνια χωριστεί από ένα τείχος. Στην Ιερουσαλήμ υπάρχει ένα αντίστοιχο τείχος. Τέτοιες ιστορίες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό είναι για αυτό το λόγο είναι υποχρέωση μας να δράσουμε. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Ζήμερ. Ε, όπως ξέρετε κυρία Ζολή, στην ε, Ιερουσαλήμ συναντήσαμε και έναν Ισραηλινό, έναν Εβραίο που μιλούσε για ένα μέρος, για ένα τμήμα του λαού του, λέγοντας ότι είναι πονίδιστη η πράξη της κυβέρνησης του Ισραήλ, ε, εξέφρασε τη λύπη του και γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι οι Ισραηλινοί δεν δέχονται αυτή την απόφαση και αυτή την πορεία. Και έχουμε να, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση είναι οδυνηρή και για αρκετούς ε, Ισραηλινούς. Έχετε το λόγο. Όλοι. Ε, ε, Νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία έτσι ώστε το θέμα να διασαφινιστεί πλήρως. Να επεξηγήσουμε τα γεγονότα και οι Ισραηλινές αρχές να δώσουν μια επεξήγηση στη ε, κοινή γνώμη, στη διεθνή κοινή γνώμη. Νομίζω ότι ο ρόλος της Ευρώπης ε, θα πρέπει να αφορά μια διαδικασία, μια διαδικασία ειρήνευσης, έτσι ώστε όλοι να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι για να μιλάμε για ευθύνες οι οποίες επιμερίζονται. Η Ευρώπη είναι η μεγάλη απούσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εδώ και πολύ καιρό, ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαίοι ε, ανακαλύπτουν ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και εκφράζουν τη λύπη τους. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ήμασταν ε, απόντες. Νομίζω, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Μίτσελ, το να καλέσουμε και την Αίγυπτο είναι πολύ σωστό, αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Διότι η κατάσταση της Γάζας αφορά και ευθύνες της Αιγύπτου. Μιλάμε για μία ε, λωρίδα, μία μικρή λωρίδα την οποία δεν θέλησε κανένας. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει ένας διάλογος. Θα ήθελα να καλέσουμε τον Τόνι Μπλερ να μας επεξηγήσει τι συνέβη με την αποστολή του στη Μέση Ανατολή. Διαφορετικά, την επόμενη φορά θα, ξε... θα ξυπνήσουμε διαπιστώνοντας εκ νέου την ανικανότητά μας και δυστυχώς θα προκύψουν και νέες στρατιωτικές δραστηριότητες. Ευχαριστούμε. Ήδη έχει γίνει ακρόαση του Τόνι Μπλερ στην Επιτροπή μας και ε, θα πρέπει να πω ότι δεν εντυπωσιάστηκα από αυτά που είχε να μας πει ε, για την αποστολή του ως προς την επίλυση της ε, λύσης. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, Νομίζω ότι η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια φέρει μεγάλη ευθύνη για την απουσία της. Όταν εκφραστούν όλοι, να ανακεφαλαιώσουμε την κατάσταση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ. Έχουμε να κάνουμε με μία μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία, είναι σαν να έχουμε τον Άμλετ χωρίς τον ε, πρίγκιπα της Δανημαρκίας. Εμείς ε, επικουρήσαμε με ευρώ αυτή την ε, ανθρώπινη, ανθρωπιστική τραγωδία και τίποτα δεν έχει αλλάξει διότι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δυσκολίες, δαπανά πολλά χρώματα, χρήματα συγγνώμη, από τον συρρυκνούμενο προϋπολογισμό της για να αντιμετωπίσει την κατάσταση των προσφύγων τη στιγμή που οι γείτονες αραβικές χώρες που είναι ιδιαίτερα πλούσιες που έχουν πολλά, διαθέτουν πολλά χρήματα δεν ενδιαφέρονται καν για την πρόνοια των ε, συναδέλφων των, των μουσουλμάνων φίλων. Είναι πολύ επώδυνο για αυτούς. Και πρέπει να γίνει σημαντικό και για τις γείτονες χώρες, δηλαδή να καταλάβουν ότι θα πρέπει να ενισχύσουν ε, την ασφάλεια και των δύο πλευρών και του Ισραήλ. Διαφορετικά δεν θα καταλήξουμε πουθενά αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό. Τη στιγμή μεγάλων χρηματοοικονομικών δυσκολιών, δεν, γιατί δεν ζητάμε από τα αραβικά κράτη να αναλάβουν αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος υποβάλλει αυτή την ερώτηση, είναι επώδυνο βέβαια. Αλλά μόνο όταν προωθηθεί κάτι τέτοιο, τότε θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και των δύο κοινοτήτων. Διαφορετικά, αν δεν γίνει τίποτα στο Ντουμπάι, στο Ριάντ ή οπουδήποτε άλλο στα ε, αραβικά κράτη, στο Κατάρ, οπουδήποτε άλλο, τίποτα δεν θα συμβεί. Και θα μας γελιοποιήσουν. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν στην ουσία. Θα πρέπει εμείς να προωθήσουμε αυτό το διάβημα στα αραβικά κράτη να αναλάβουν την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια προς, τα, προς Παλαιστινίους που έχουμε αναλάβει εμείς. Και αν αρνηθούν θα ξέρουμε πώς να συνεχίσουμε. Madame Κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η η κατάσταση στη Δυτική Όχθη είναι εντελώς διαφορετική από την κατάσταση στη Γάζα. Δεν είναι δυνατό να κάνουμε σύγκριση ανάμεσα στα δύο. Στη Γάζα, εκτός από τον φρικτό αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ, υπάρχει και μια ιδιάζουσα κοινωνική διαφοροποίηση λόγω των κλειστών γάμων που επιτελούνται στην περιοχή αυτή. Πρώτα ξαδέρφια, ακόμη και αδέλφια παντρεύονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές συγγενείς ανομαλίες, συγγενείς διαμαρτίες στα παιδιά που γεννιούνται και αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα. Πέρα από την απόλυτη φτώχεια μέσα στην οποία όπως πολύ σωστά μας έχει δει εκπρόσωπος της ΟΥΡΑ ζουν ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό του πληθυσμού και την καταστροφή της οποιασδήποτε υποδομής δημιουργείται. Κάθε λίγο και λιγάκι με τους βομβαρδισμούς καταστρέφεται οποιαδήποτε υποδομή προσπαθεί να δημιουργηθεί από τον λαό. Μας μιλήσατε για αρκετές χιλιάδες τούνελ τα οποία υπάρχουν και με τα οποία μπαίνει υλικό. Υποθέτω ότι αυτά τα τούνελ είναι στα, κοντά στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίπτο, διότι στη Δυτική Όχθη δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Και το ερώτημα είναι, αντιλαμβάνεται κανένα την ευθύνη της Αιγύπτου που δεν επέτρεπε. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, που ασκεί κρατική τρομοκρατία και συνεπώς δεν, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο μπορεί η διεθνής κοινότητα να διαφοροποιήσει τη συμπεριφορά του. Εκτός από αυξημένες κυρώσεις που δεν είναι κανένας διατεθειμένος να τις επιβάλλει. Η Αίγυπτος δεν είχε υποχρέωση όλα αυτά τα χρόνια να ανοίξει τη ράφα για να μπορεί να τροφοδοτείται η Γάζα. Ένα ερώτημα βασικό. Δεύτερο, το Ισραήλ ναι, αλλά το έκανε χτες. Το Ισραήλ ισχυρίστηκε χτες με τον ε, ε, πρέσβη του, τον εξοχότατο που ήρθε και μας μίλησε στην Επιτροπή Εξωτερικών, ότι γίνεται διείσδυση όπλων προς τη Γάζα από καράβια. Και το ερώτημα που δεν απάντησε ποτέ είναι γιατί δεν έπιασαν ποτέ ένα τέτοιο καράβι και πάντα επιτίθενται εναντίον αόπλων ακτιβιστών. Και αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί ήμουν πάνω στον Τίγνητη στις 29 του Δεκέμβρη όταν μας επιτέθηκε το ναυτικό, εμβόλισε το πλοίο και παρολίγο να μας πνίξουν και μας έσωσε το γαλλικό ναυτικό. Συνεπώς όλες αυτές τις ψευτιές και τις ε, δεν μπορεί να τις πουλούν σε Ευρωπαίου. Ε, ευρωβουλευτές. Είναι γι' αυτό το λόγο που εκείνες τις μέρες αμέσως μετά τη βήθηση του Dignity η κυρία Μπακογιάννη, Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, είχε ζητήσει το άνοιγμα ενός διάβλου, θαλάσσιου διάβλου, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά της Κύπρου και της Γάζας, για να διασωθεί ο πληθυσμός. Είχε πάρθει μία απόφαση. Ξεχάστηκε και το dignity, ξεχάστηκε και η βήθησή του, ξεχάστηκαν όλα. Και αυτά που συμβαίνουν σήμερα θα ξεχαστούν σε 15-20 μέρε. Ο λαό τη Γάζα όμω θα είναι εκεί και θα υποφέρει. Και δεν μπορεί μόνο με τι θεωρίε μα και τι αναλύσει μα και τι θεωρητικέ προσεγγίσει να αφήσουμε να εξελίσσεται αυτό το δράμα. Χτε πάλι, έχω τον χρόνο, ε, κυρία Πρόεδρε. Nous sommes terriblement en retard. Έχουμε αργοπορήσει πάρα πολύ. Έχουμε άλλο ένα σημείο στη μερίσια διάταξη και πρέπει να κλείσουμε. Όλοι συμφωνούμε. Είναι τραγική η κατάσταση. Το σημαντικό είναι να αφιερώσουμε επαρκή χρόνο τόσο ώστε να αποφασίσουμε για τη μελλοντική μας δράση. Θα, θα, θα καταλήξω λέγοντας ότι είναι αδύνατο για τη διεθνή κοινότητα να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει στη Γάζα, αλλά αν δεν πάει και να ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους για λίγο καιρό. Και το βασικό ερώτημα, η Χαμάς τι προσφέρει και έχει ένα τόσο υψηλό ποσοστό ε, ψήφων. Ήμουνα, ε, έκανα τον, το, το monitoring των εκλογών και ήταν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο που κέρδισε η Χαμάς. Έτσι γιατί δεν σκεφτόμαστε τι είναι εκείνο που κάνει του Παλαιστίνιου να ψηφίσουν τη Χαμά. Μια τρομοκρατική οργάνωση. Όπω έχω πει ότι το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκράτη, το ίδιο λέω και για την Χαμά. Γιατί, γιατί του δίνει ψωμί και τρώνε όταν δεν έχουν τίποτε άλλο. Ευχαριστώ κατάσταση αυτή ε, συνεχίζεται εδώ και 60 χρόνια ανάμεσα στην Παλαιστίνη και ιδιαίτερα στη Γάζα ε, και το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι ε, τώρα επαναλαμβάνοντας αυτά τα πράγματα. Ε, μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που συνέβη στα διεθνή χωρικά ύδατα αυτή τη βδομάδα, να επιμείνουμε να εκπονηθεί διεθνή έκθεση, ε, γιατί είναι ένα γεγονός και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι έχουμε μια ευκαιρία να σημειώσουμε πρόοδο. Εάν διεξαχθεί δε η μελέτη από ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες, θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο κάποιας μελλοντική δράσης, διότι μπορεί η έκθεση να στοιχειοθετήσει την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, του δικαίου του πολέμου. Ας εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή μας σε αυτό το συγκεκριμένο μεμονωμένο γεγονός για να σημειώσουμε πρόοδο. Αυτό που με ανησυχεί είναι το ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχει αποφασίσει να ζητήσει την διεξαγωγή της μελέτης αυτής. Και άρα σε αυτό έγκυται κατ' εμέ η ευθύνη της Ευρώπης. Σήμερα εμείς πρέπει να ζητήσουμε ε, την ε, παρέμβαση διεθνών αμερόληπτων εμπειρογνωμόνων αυτή την ευθύνη πρέπει να υπομειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ψηφίσματος, κατά τη γνώμη μου, ή και μέσω σύστασης προς το Συμβούλιο. Η σύσταση προς το Συμβούλιο μπορεί να γίνει από τις πολιτικές ομάδες ή από 40 βουλευτές. Δεν είμαστε αρκετοί λοιπόν εδώ στην Επιτροπή ανάπτυξη για να συντάξουμε αυτή την σύσταση προς το Συμβούλιο. Ο καθένας από εμά στην πολιτική του ομάδα μπορεί να εργαστεί για αυτό, για να υπάρξει υποστηρίξη ούτω ώστε να γίνει σύσταση προς το Συμβούλιο να ζητήθει εξωτερική αμερόληπτη εμπειρογνωμοσύνη, τεχνογνωσία. Πρέπει να διοριστεί ένας εμπειρογνώμονας. Εάν δεν γίνει αυτό από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μπορεί ενδεχομένως να διοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μετέλθει των μέσων του λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπερψηφίσει ένα ψήφισμα στην επόμενη Ολομέλεια για αυτό το θέμα. Αυτή είναι η εισήγηση που σας κάνω. Βέβαια μπορούμε να ε, ε, εκπονήσουμε και, μια, και ένα πληρέστερο ψήφισμα, όπως είπε ο κύριος Γκέι Μίτσελ, ε, να επιδιώξουμε τη δίωδο μέσω Αιγύπτου ε, με μέσα που δεν περιορίζονται σε αυτά που αυθαίρετα αποφάσαν οι Ισραηλίν, να ε, αφήνουν να περνούν εν είδη ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτά λοιπόν συνοψίζοντας να επικεντρωθούμε σε αυτά που έγιναν στα διεθνή χωρικά ύδατα και να επιμείνουμε για τη μελέτη. Αν ε, ε, το πόρισμα της μελέτης είναι ότι υπήρξε παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι αυτή περιπτώσει υπάρχουν διεθνείς δικαιοδοτικές αρχές που μπορούν να δικάσουν τους αξιωματούχους που έδωσαν τις εντολές. Άρα θα υπάρχουν νομικές συνέπειες στη συνέχεια. Ο κύριος Σασόλη. Θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δύσκολο να λάβει πρωτοβουλίες γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Ισραήλ προβαίνει σε μία ε, κρατική τρομοκρατία. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη. Θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να βρούμε το σωστό τρόπο για να διαβιώσουν οι άνθρωποι ειρηνικά. Ε, επιβεβαιώνοντας την, ε, και υπενθυμίζοντας την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ότι θα πρέπει να καταστέλλονται οι παραβιάσεις, αλλά μιλάμε και για μια κατάσταση έκριθμη Δεν θα θέλαμε το Ισραήλ να αποτελεί παράδειγμα, γιατί υπάρχουν υπάρχουν και υπάρχει και η δυνατότητα για τους πολίτες να αλλάξουν γενικότερα πολιτική. Ε, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μαζί με, εκείνον, με που σκέφτονται το θέμα μόνο μονομερός και θεωρούν ότι μπορεί να επιληθεί ε, μόνο ε, με δράση κατά του Ισραήλ. Τρία ζητήματα εθίγησαν από την Πρόεδρο θα ήθελα να υποστηρίξω τους κύριους Κάσμαν και Τζίμερ που μίλησαν για ένα ψήφισμα για την σύνταξη ενός ψηφίσματος έτσι ώστε να εφαρμοστεί το άρθρο 2, δηλαδή η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την άρση συνεργασίας με το Ισραήλ. Και τα αραβικά ε, κράτη όμως θα πρέπει να διαδραματίσουν το σωστό ρόλο. Δεν μπορούμε να το διευθετήσουμε τώρα. Νομίζω ότι θα ήταν ε, σκόπιμο να δούμε τι συνέβη και αν θέλουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να δούμε τι ρόλο θα ε, διαδραματίσουμε εμείς σήμερα Ίσως χρειαστούν και 30 χρόνια για να διευθετούν τα υπόλοιπα Μίτσελ. Υποστηρίζω αυτά που είπατε. Δεν μπορούμε να το επιλύσουμε ολιστικά την μεθεπόμενη εβδομάδα θα είμαστε στο Στρασβούργο. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και η διάσκεψη των Προέδρων και μέχρι τότε θα αποφασίσουμε πώς θα το χειριστούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τώρα, αλλά την μεθεπόμενη εβδομάδα οπωσδήποτε θα μας ενημερώσει η Βαρονή Άστον. Αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει εδώ και τώρα. Ο κύριος Κέρενς, Συμφωνώ απόλυτα κατά με τον ε, κύριο Σασόλη, αν και ε, ανήκουμε σε διαφορετικές ομάδες. Το Ισραήλ είναι μια χώρα τρομοκρατών. Δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ε, ακολουθούμε τόσο παθιασμένη αντιμετώπιση. Εντάξει, ωραία, θα πρέπει να υπάρξουν δύο κράτη σίγουρα, αλλά με μεγαλύτερη ε, ηρεμία θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Να δούμε πώς ε, διατραματίστηκαν τα γεγονότα. Πριν κρίνουμε θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα. Ελπίζω να γίνει μια διεθνής έρευνα και στη συνέχεια θα αποσαφινιστεί το όλο ζήτημα. Μάλιστα κύριε Γκέρενς, ευχαριστώ πρόεδρε. Η μακρά παράδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας δείχνει ότι όλα τα ψηφίσματα, σχεδόν όλα, ε, ε, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Οπότε αν κάνουμε μία μακροσκελέστατη τέτοια πρόταση με 36 συστάσεις και 72 σκέψεις, τίποτα δεν θα καταφέρουμε. Σας το εγγυώμαι. Δύο είναι οι διαστάσεις της μελλοντική δράσης του Κοινοβουλίου, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, όπως είπατε, εσείς πρόεδρε, χρειάζεται διεθνής έρευνα, γιατί υπάρχει υποστήριξη και στο Ισραήλ για αυτό. Ε, αυτό συνέβη σε διεθνή χωρικά ύδατα, εάν ε, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να διεξάγουμε διεθνή μελέτη, δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Δεύτερη διάσταση. Η Ούνβρα έχει αρμοδιότητα για να δράσει επιτόπου στη Γάζα, αλλά δεν έχει ελευθερία κινήσεων. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και αυτό παραβιάζει την αρχή της αμεροληψίας σε κάθε ανθρωπιστικής παρέμβασης, είτε μιλάμε για θεσμική είτε για διεθνή παρέμβαση. Πρόκειται για ένα θεσμικό εταίρο που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει να αφήσουμε την Ούντρα να κάνει τη δουλειά της. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποδεέστερα και μας αποτρέπουν από τον πολιτικό μας στόχο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βιλάρ και πάλι τώρα για να απαντήσει στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Ευχαριστώ κυρία Ζολή. Ευχαριστώ κύριε Γκέρενς για την υποστήριξή σας για το έργο της ΟΝΡΑ στη Γάζα. First of all, thank you to... Να ευχαριστήσω και την κυρία Κρετού, η οποία δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, για την υποστήριξη των δράσεων μας στη Γάζα και την αντιπροσωπεία για το αίτημα που εξέφρασε για την οικονομική ενίσχυση για να συνεχιστούν οι δραστηριότητες μας όχι μόνο στη Γάζα αλλά και σε άλλους πέντε τομείς. Όπως είπα, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, μια πολύ σοβαρή οικονομική κατάσταση, το πιο σοβαρό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ποτέ. Ε, δεν υπάρχει καν η παροχή ε, βασικών ε, υπηρεσιών. Μιλούμε για 73 εκατομμύρια ευρώ από έναν προπολογισμό 428 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Ονρα δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της μετά το Σεπτέμβρη, εάν η κατάσταση συνεχίσει να είναι αυτή που είναι. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιο έλλειμμα, τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά. Και γι' αυτό ζητούμε ενίσχυση, υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή είναι η βασική μας, ο βασικός μας υποστηρικτής και τα κρατημέλη και η Κομισιόν. Και έχουμε πάρα πολύ δραστήρια, συνεχή αιτήματα για οικονομική βοήθεια. Έχουν γίνει προσπάθειες και για την βοήθεια από τις αραβικές χώρες για να ξεκαθαρίσουμε για τη δική τους ε, ενίσχυση, έχετε δίκιο κύριε Ντέβα και η κυρία Κρετού επίσης, ότι συμβάλλουν μόλις 1,5% στο γενικό ταμείο της Ούνρα οι αραβικές χώρες. Αυτό είναι ένα τμήμα του προπολογισμού μας. Είναι ε, έτσι όπω πληρώνουμε τους ε, μισθού των γιατρών, των δασκάλων. Αυτό είναι ο, προπολογισμό για τον οποίο σας μίλησα ε, πριν, για τα 428 εκατομμύρια δηλαδή. Αυτοί συμβάλλουν κατά 1,5%. Υπάρχει λοιπόν μια, ένωση, μια, υπάρχει μια δήλωση από την Αραβική Ένωση ότι θα συμβάλλουν κατά 7,8%. Πιέζουμε όσο είναι δυνατόν και ο Γενικό Επίτροπο ήταν εκεί στη Σαουδική Αραβία την προηγούμενη εβδομάδα και προσπαθούμε να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους άραβε δωρητέ, και πρέπει να πω ότι υπάρχει και άλλο ένα τμήμα του προπολογισμού μας που περιλαμβάνει ε, ad hoc προγράμματα, επίγοντα αιτήματα, ε, κοινωνική, δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας ας πούμε, όπου καλύπτονται οι πιο φτωχοί. Οι αραβικές χώρες συμβάλλουν σε αυτά τα επίγοντα αιτήματα και σε αυτά τα προγράμματα. Συμβαίνει αυτό και μάλιστα συμβάλλουν και, ένα, σε ένα σημαντικό ποσοστό. Οπότε σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε μαζί σας ότι όντως πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για να λάβουμε επιπλέον ε, ενίσχυση από τις χώρες ε, τις αραβικές, αλλά ήδη συμβάλλουν όχι στο γενικό μας προπολογισμό, αλλά σε άλλα προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, Έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα κονδύλια από τις αραβικές χώρες, γιατί πραγματικά είναι καλοδεχούμενα. Merci Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εργασία αυτή, για την εξαιρετική εργασία και τις προσπάθειές σας στη Γάζα. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι τα μέλη των τριών επιτροπών που ε, παρευρέθησαν, βρέθηκαν στη Γάζα θα συντάξουν ένα κοινό ψήφισμα για την Ολομέλεια του Ιουνίου που καταγράφει αυτά που είδαμε στη Γάζα και αυτά που θεωρούμε ενδεδειγμένα για να βρούμε μια λύση. Οι τρεις γραμματείες αυτών των επιτροπών, ΑΦΕΤ, ΔΕΒΕ και Μπάτζετ, είναι επιφορτισμένες ε, με τη σύνταξη του σχεδίου του ψηφίσματος υπό τον έλεγχο των βουλευτών που ήταν επιτόπου. Ελπίζω να συμφωνείτε με το διάβημα για το ψήφισμα για την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα. Αυτό δεν ρυθμίζει βέβαια το πρόβλημά μας για το ενδεχόμενο αίτημα για διορισμό διεθνών ανεξαρτήτων εμπειρογνωμών. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω υπό ποια μορφή, υπό, με ποια διατύπωση, ποια διατύπωση θα έχει το αίτημα. Δηλαδή, σύσταση θα είναι προς το Συμβούλιο, ψήφισμα, θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Μπορούμε να παραμείνουμε σε επαφή ε, με όσους ε, είναι επιφορτισμένοι με τη σύνταξη του σχεδίου ή να φτιάξουμε μια μικρή ομάδα εργασίας για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα για το διορισμό των ε, ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων. Ο κύριος Γκέρενς. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Υποστηρίζω αυτή την τελευταία σας πρόταση. Λοιπόν, ε, συμφωνήσαμε επί δύο σημείων. Νομίζω υπάρχει συνένεση, διεθνή έρευνα δηλαδή αφενό, αφετέρου να επιτρέψουμε στην Ούνρα να κάνει τη δουλειά τη ε, υπό μορφή συστάσεων ε, βάσει του άρθρου 121 του καταστατικού μα. Έτσι, εγώ προτείνω σύσταση προ το Συμβούλιο. Από τότε που κάναμε τη συζήτηση, είχαμε και μια συνάντηση συντονιστών ε, μάλλον θα έχουμε και μια σε μια ε, συνάντηση συντονιστών, οπότε ας το σκεφτούμε και ας το συζητήσουμε και εκεί. Έχουμε και ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Δύο ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δείτε τα ερωτήματα στο φάκελό σας. Μόνο ο βουλευτής που έχει συντάξει την ερώτηση μπορεί να κάνει επερώτηση. σα το υπενθυμίζω. Η κυρία Κέλλερ και ο κύριος Μπέγκμαν έχουν συντάξει την πρώτη ερώτηση. Δεν χρειάζεται να στη διαβάσουμε. εμεί στο φάκελό σα. Επιτροπή. της Επιτροπής θα μας δώσει την απάντηση. Παρακαλώ. Uh, yes, uh, thank you. The Commission Ευχαριστώ. Ε, με χαρά έδεχθη την ερώτηση η Κομισιόν για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα έχουμε την ε, δυνατότητα να ε, εξηγήσουμε τώρα το τι ακριβώς κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά ε, ώστε να βοηθήσουμε την πρόσβαση σε πολιτιστικά προϊόντα για άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, οικομισιών μαζί με τα κράτη-μέλη. Και είναι αλήθεια ότι στην επόμενη μόνιμη επιτροπή τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν καταφέρουμε να λάβουμε την ευλογία της, θα προτείνει μία σύσταση η οποία θα είναι πολύ λεπτομερής και θα περιλαμβάνει τις συστάσεις που όλες θα πρέπει να έχουν φροντίσει να έχουν εξαιρέσει οι χώρες μέλη για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Γιατί αυτό στο πρωτογενές δίκαιο και όχι στη συνθήκη που είναι, που είναι κάτι που έχει ε, υποστηρίξει η Παγκόσμια Οργάνωση Τυφλών με υποστηρίξη Βραζιλίας και Νικαράγουα. Το κάνουμε αυτό γιατί είναι πιο γρήγορο. Είναι αποτελεσματικό, εφαρμόζεται άμεσα. Η συνθήκη θέλει πολλές διαπραγματεύσεις και μετά από τις πολλές διαπραγματεύσεις πολλές χώρες θα πρέπει να την επικυρώσουν πριν αρχίσει να εφαρμόζεται, πριν τεθεί σε ισχύ. Ε, υπάρχουν πολλές ε, συνθήκες WIPO ε, που, πρέπει που συνήθως χρειάζονται 50-60 χώρες να τις επικυρώσουν για να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ. Επίσης θα πρέπει να αλλάζαμε την, ε, το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν ε, διεθνείς συνθήκες που ήδη περιλαμβάνουν εξαιρεσει. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει εξαιρεσει για τα άτομα με αναπηρία, και καμία από αυτές δεν είναι υποχρεωτική. Αλλά όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, προβλέψει κάτι για, τα, για τους πολίτες με ε, προβλήματα όραση. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα λοιπόν, ένας διάλογο ε, με εκπροσώπου από το Φόρουμ για το Άτομα με Αναπηρία και από την Παγκόσμια Οργάνωση ε, Τυφλών. Ε, αυτή είναι μια προσέγγιση άμεση που την ξεκινήσαμε πριν από τη Μόνιμη Επιτροπή, ήδη από πέρσι το Δεκέμβρη. Αυτό ο διάλογο λοιπόν μελετά συγκεκριμένα την αύξηση στην παραγωγή ε, προϊόντων ε, σε προσβάσιμη μορφή σε όλη την Ευρώπη. Ε, θέματα τεχνολογίας, ε, διαλειτουργικότητα όλων αυτών των φορμάτ που υπάρχουν με όλες τις συσκευές που πρέπει να χρησιμοποιούν ε, τα άτομα με αναπηρία. Επίσης προσπαθούμε να, να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει κοινοποίηση για το πού βρίσκονται αυτές οι προσβάσιμες, αυτά τα προσβάσιμα format, πώς μπορεί κανείς να καταχωρηθεί και να έχει πρόσβαση σε αυτά ως άτομο με αναπηρία ή τυφλός. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης, πολύ άμεσο, θα γίνει ένα μνημόνιο κατανόηση για όλα αυτά, το οποίο θα υπογραφεί στι 30 Ιουνίου. Θα γίνει μια αξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο λειτουργεί. Η WIPO έχει έναν διάλογο επίση, ο οποίο ε, είναι σε εξέλιξη εδώ και κανένα δύο χρόνια για, και θα συνεχιστεί για ένα-δύο χρόνια ακόμη, που επίσης μελετά θέματα τεχνολογία και θέματα διαλειτουργικότητας και βάση δεδομένων. Και νομίζω ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία θα μπορέσει να είναι χρήσιμη για τον διάλογο του WIPO πολύ πρακτικά και αρκετά αποτελεσματικά θέλω να πιστεύω. Θα καθοριστούν κανόνες για τους, ε, εμπιστευ... για τους ε, ε, που χαίρουν εμπιστοσύνη, γιατί υπάρχουν ήδη τέτοιες οργανωμένες δράσεις και ελπίζω να τους έχουμε σε όλα τα 27, και στα 27 κράτη-μέλη και ο διάλογος επίσης θέλει να δημιουργήσει τέτοιου είδους ενδιάμεσους σε όλα τα και στα 185 κράτη, γιατί μόνο μέσω αυτών των ενδιαμέσων θα μπορέσουμε αυτοί θα μπορέσουν αυτοί που παράγουν τέτοια προσβάσιμα format ε, να ξέρουν ότι θα πηγαίνουν όντως, θα καταλήγουν στα σωστά χέρια τα προϊόντα αυτά. Υπάρχει και μια πολιτική βεβαίω πτυχή τα ευρωπαϊκά θεωρούν ότι η διεθνή νομοθεσία και οι συνθήκε ήδη συμπεριλαμβάνουν εξαιρέσει και περιορισμού και για τα άτομα με αναπηρία και για τα άτομα με προβλήματα όραση. Και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια ομάδα κρατών στη Γουάϊπο που ισχυρίζεται μάλλον αρνείται την συνθήκη που προτείνεται για τα άτομα με προβλήματα όρασης, γιατί θέλουν, άτομα, θέλουν μια συνθήκη με πιο ευρείες εξαιρέσει. θέλουν εξαιρέσει για την ε, εκπαίδευση κτλ. Ε, θέλουν λοιπόν μια μεγάλη συνθήκη γεμάτη εξαιρέσει. Αν δείτε το διεθνές δίκαιο, έχει αυτό το ε, τεστ σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει και συγκεκριμένες εξαιρέσεις Οπότε νομίζω ότι, νομίζω ότι θα, θα πάμε πολύ μακριά, θα ξεπεράσουμε τα, του... τα θέματα που έρχονται του copyright. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τους ε, δημιουργικούς ανθρώπους. Ε, μου είπατε να είμαι σύντομη, ελπίζω να μην μακρηγόρησα πολύ, αλλά θέλω να σας ε, ε επιβεβαιώσω ότι δεν είμαστε μακροπρόθεσμα κατά, ενάντια της συνθήκης, αλλά θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αποτελεσματικοί και με την τεχνική βοήθεια της WIPO να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες που τώρα ε, εισάγουν στην νομοθεσία τους νομοθεσία για το copyright, να μπορέσουμε να, ε, να δράσουμε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλέ χώρε που κάθε χρόνο ενσωματώνουν στην νομοθεσία του τέτοια νομοθεσία για το copyright με διάφορε εξαιρέσει. Ευχαριστώ. Δεν θα υποβάλω και εγώ ερώτηση, θα το κάνω την επόμενη φορά, διότι έχουμε ε, υπερβεί το χρόνο μας. La follow-up question est vraiment indispensable. Πρέπει οπωσδήποτε να ρωτήσετε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πια διερμηνία.